Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σας ε, καλωσορίζω στην ε, συνεδρίασή μας. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Δεν βλέπω καμία αντιρρήση, οπότε εγκρίνεται. Και επίση, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνονται και τα πρακτικά τη 25η και 26η Απριλίου και της 12ης και 23ης Τετάρτης και 24ης Μαΐου. Και εδώ πέρα βλέπω καμία αντίρρηση. Ωραία. Ανακοινώσει του Προέδρου δεν υπάρχει τίποτα. Και περνάμε στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Η συγκίτρια έχει το λόγο, η Μάισνερ. Να ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και καλή μέρα σε όλους τα επαγγελματικά προσόντα στην ιστορική ναυσιπλοεία ακούγεται ένα, ως ένα πολύ τεχνικό θέμα αλλά νομίζω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μετακινήσουμε κάποια κίνηση στην ιστορική νευσιπλοεία, να φύγει από τους δρόμους, να μην πάει μόνο στους σιδηροδρόμους, αλλά και στα ποτάμια. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε καταρτισμένο προσωπικό. Και υπάρχει μια έλλειψη λοιπόν, δηλαδή τα πληρώματα είναι κάπως ηλικιωμένα και δεν μοιάζει και αρκετά ελκυστικό το επάγγελμα. Δεν τρέχει ο κόσμος να απασχοληθεί εκεί πέρα. Γι' αυτό ακριβώς ασχολούμαστε και με αυτή την πρόταση. Στο πλαίσιο έτσι, της κινητικότητας των εργαζομένων έχει νόημα να μπορεί κανείς να εκπαιδευτεί σε ένα κράτος μέλος και να πάει στα ποτάμια ενός άλλου κράτους μέλους. Βεβαίως πρέπει να ξέρουμε να δούμε ποια, πότα πρέπει να ξέρει βεβαίως και τις σχετικές δυσκολίες του κάθε ποταμού αλλά νομίζω πως ε, θα πρέπει να υπάρχουν οι βασικές γνώσεις για να μπορεί κανείς να κάνει αυτή τη δουλειά σε ολόκληρη την Ευρώπη ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες βεβαίως ε, ε, είναι διαφορετικό το να μεταφέρει κανείς επικίνδυνα υλικά ή επιβάτες Βεβαίω θα ακολουθήσουν και οι συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών για να τελειώσουμε κάποια στιγμή, ελπίζω, φέτος. Αυτά. Ευχαριστώ. Όλος εξαιρετικός έχουμε και κάποιους ειδικού. Πρώτα απ' όλα την ε, κυρία Τέρεζα Χακστάινερ από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Λάντζων και σχετικών πλοίων. Uh, um, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που καλέσατε την EBU στη σημερινή σας συνεδρίαση. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τη δική μας άποψη για την πρόταση αυτή. Όπως είπε και η κυρία Μάσινερ, είναι όντως πολύ σημαντική πρόταση και για τον κλάδο. Η EBU ε, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους στους, στις Λάντζες και τα συναφή πλοιάρια. Ε, αυτή η πρόταση ε, ακολουθεί μια πρωτοβουλία της ε, EBU ήδη από το 2004, όπου είχαμε ζητήσει μια εναρμόνιση των προσόντων ακριβώς για τους λόγους που τόνισε και η εισηγήτρια. Λόγω της έλλειψης καταρτισμένων προσώπων στον κλάδο αυτό, και για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την, ε, ένα υψηλό πρότυπο ασφάλειας, είχαμε ζητήσει αυτή την αρμόνιση. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτή την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και στα πλαίσια αυτής της ε, νέας πρότασης, που θέλει να διευκολύνει την καλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη, και να δημιουργήσει ένα σύστημα μεικτής αρμοδιότητας ε, παρά ένα σύστημα που θα βασίζεται στην κατάρτιση θα πρέπει να προσελκύσει νέους αλλά και ε, άτομα που βρίσκονται εκτός του κλάδου. Και νομίζω ότι με το σύστημα αυτό, ε, με, την εναρμόνιση των προσόντων και την αναγνώριση, νομίζω ότι αυτό το σύστημα θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και να προσελκύσει αυτά τα άτομα. Τώρα για τα πρότυπα πρέπει να τονίσουμε ότι για την EBU θεωρείται η ναυσιπλοεία ως ο πιο ασφαλής ε, τρόπος μεταφοράς και βεβαίως πρέπει να διατηρηθούν τα πρότυπα που υπάρχουν ειδικά όταν πρόκειται για μεταφορά επικίνδυνων υλικών στην ε, Ευρώπη. Ένας από τους πιο σημαντικούς ε, τρόπους για να μεταφερθούν τέτοιου είδους υλικά είναι ακριβώς η θαλάσσια οδός ή η ναυσιπλοεία εσωτερική. Και Βεβαίως πρέπει να φροντίσουμε τα αντίστοιχα πρότυπα για τη μεταφορά επιβατών. Τονίζουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πρότυπο μετά από στενή συνεργασία με όσους έχουν την εμπειρία στον τομέα αυτό και αναφέρομαι στην Επιτροπή ΣΕΣΝΗ που δημιουργήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της CCNR, της Επιτροπής του Ρήνου, για να ασχοληθεί και με την τεχνική, και με την πρόταση αυτή, αλλά και με την τεχνική οδηγία η οποία έχει υιοθετηθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Και σύμφωνα με, τούτε στις, με την προσέγγιση, είναι καλό να υπάρχει ε, το σύστημα αυτό προσόντων, το οποίο θα ελέγχεται από τους εμπειρογνώμονες στον κλάδο και βεβαίως θα εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εμπειρογνώμονες του κλάδου. Είναι σημαντικό αυτό για ε, εμάς να μην ε, αποδυναμωθούν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα. Τώρα, άλλη μια ανησυχία που απασχολεί τον ε, κλάδο είναι το θέμα της αποφυγής του certification shopping. Να διατηρήσουμε δηλαδή τα πολύ αυστηρά πρότυπα ασφάλειας που έχουμε μέχρι τώρα και θα πρέπει να αποφύγουμε την έκδοση πιστοποιητικών από τα κράτη-μέλη τα οποία ίσως να μην είναι εξοικειωμένα με την εκπαίδευση, με την κατάρτιση για την αυσιπλοεία. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί. Τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, τέτοιες οδούς ε, ναυσιπλοείας να μην μπορούν να εκδίδουν ε, τέτοιου είδους πιστοποιητικά για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι το πρότυπο ασφαλείας θα παραμείνει υψηλό. Κλείνοντας, για να διαφυλάξουμε αυτά τα δύο βασικά στοιχεία, Καλωσορίζουμε την πρόταση αυτή, αλλά ταυτόχρονα ζητούμε και από τα εμπλεκόμενα μέρη να εγγυηθούν την ε, ασφάλεια σε στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Την ε, Επιτροπή του Ρήνου, της ΕΣΕΝΑΡ δηλαδή κυρίως, που έχει την εμπειρογνωμοσύνη μέσω της ΣΕΣΝΗ, την Επιτροπή που δημιουργήθηκε για να καθορίζει τα πρότυπα αυτά, τα οποία θα μπορέσουν να εγγυηθούν την ύπαρξη ψηλών αυστηρών προτύπων Κάτι που ούτω ή άλλω είναι και ο στόχο αυτή τη πρόταση. Και επίση, όπω είπα, σε, το, στο βαθμό που μπορούμε να αποφύγουμε το certification shopping. Ευχαριστώ. Η κυρία Μίριαμ Σαφάρ από την ε, Ένωση Ευρωπαίων ε, Εργαζομένων στις Μεταφορές. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ε, δικής μας νομοσπονδίας. θα ήθελα να ε, σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου που, ακούσατε τις, ε, που θα ακούσετε τις απόψεις μου. Ήδη η, η TWF καλωσορίζει την πρόταση αυτή. Προκύπτει μετά από πολλά χρόνια στενή συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τον, την Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Εργαζόμενων και εργαζομενων κυβερνήσει, κυβερνήσεις, ε, ε, κέντρα κατάρτισης, κράτη-μέλη. Όπως ξέρετε όλοι, ο τομέας της εσωτερικής ναυσιπλοείας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και κυρίως δημογραφικές προκλήσεις. Η μέση ηλικία των ε, καπετάνιων είναι περίπου 50 και σε κάποιες περιοχές ξεπερνά και τα 55 έτη. Επίσης θα ξέρετε ότι ο όγκος των εμπορικών φορτίων αυξάνεται στην Ευρώπη και επίσης υπάρχει μείωση στις αστεριότητες. Η ε, βιομηχανία των, ε, της εσωτερικής ναυσιπλοείας επίσης χρειάζεται ε, περίπου 4.000 έξτρα άτομα προσωπικό για να μπορέσει να επανδρώσει τα πλοία. Και επίσης η εσωτερική ναυσιπλοεία ως, ως βιώσιμος κλάδος και φιλικό προς το περιβάλλον θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρω στην ε, ε, παγκόσμια αλυσίδα ε, για να μπορέσει να μεταφέρει μεγαλύτερο όγκο και εμπορευμάτων και επιβατών. Πρέπει λοιπόν να γίνουν διάφορες αλλαγές στον κλάδο αυτό. Ο αυτοματισμός έχει περάσει στον κλάδο Χρειάζεται όμως και εξυγχρονισμός και αυτό σημαίνει νέα προσόντα, νέες αρμοδιότητες. Για να μπορέσει ο κλάδος να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις θα πρέπει να είναι βιώσιμος και θα πρέπει να γίνει ελκυστικός. Το σεβασμός για τα μέλη των πληρωμάτων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία. Η οδηγία αυτή λοιπόν ουσιαστικά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την δημιουργία ε, ποιοτικών ε, προσόντων για τους εργαζόμενους στον κλάδο αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης θα συμβάλλει και στην διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων και θα ενισχύσει βεβαίως και την ελκυστικότητά του. Επίσης θα βάλει ένα τέλος σε παράνομες πρακτικές που ε, διακυβεύουν αυτή τη στιγμή το την κατάσταση και θα αποτελέσει ένα βήμα προς ένα πιο εξχρονισμένο κλάδο που θα παράσχει ποιοτική κατάρτιση, ποιοτική εκπαίδευση. Για την ETF, ο τελικός στόχος αυτής της οδηγίας θα πρέπει να παραμείνει να το να υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα για όλες τις ιστορικές οδούς ναυσιπλοείας χωρίς να υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα. Πρέπει να αποφύγουμε ένα διτό σύστημα και δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ ε, συνδεδεμένων ή μη ε, οδών ναυσιπλοείας. Όλα θα πρέπει να καλύπτονται από τούτη την οδηγία. Μια εναρμονισμένη οδηγία, ένα σύστημα που θα είναι εύκολο στην εφαρμογή και στον έλεγχό του αν χρειαστεί να υπάρξουν ε, εξαιρέσει ή αν υπάρξουν προβλήματα, ίσως να μπορούμε να παράσχουμε μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο στα κρατημέλη για να τους δώσουμε την ευκαιρία να εφαρμόσουν αρμοδίως την οδηγία. Σε πρώτη ανάγνωση όμως, το κείμενο της οδηγία έχει κάποιες, ε, κάποια κενά. Αν διαβάσουμε το άρθρο 2 στο προήμιο, υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος εξαιρέσεων και για εμάς η μη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία θα οδηγήσει ουσιαστικά σε νομική ασάφεια στο μέλλον. Πρέπει να ξέρουμε ότι για τις εσωτερικές οδούς ναυσιπλοείας δεν υπάρχει ε, νομοθεσία που να μιλά για το κράτος σημαίας, οπότε θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος τρόπος, ενιαία εφαρμογή της οδηγίας για να αποφύγουμε οποιοδήποτε πρόβλημα στο μέλλον. Οποιαδήποτε εξαίρεση στο άρθρο 35 είναι απαράδεκτη για μας κάθε εξαίρεση αντίκειται στον πυρήνα αυτής της οδηγίας, στον στόχο της οδηγίας, που είναι η βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν και κάποια ακόμη ίσον σημασία στοιχεία που θέλω να θίξω. Στο άρθρο 3 λέει other person, άλλα άτομα πέραν του προσωπικού που μπορεί να λάβει μέτρα σε επίγουσες καταστάσεις πάνω στα επιβατικά πλοία. Για μας αυτό το other person, άλλο άτομο, θα πρέπει να οριστεί ε, πολύ συγκεκριμένα άλλο άτομο που θα έχει κάποια καθήκοντα σε, πάνω στο πλοίο. Στο άρθρο 10 αναφέρεται ότι η μέγιστη διάρκεια ισχύω των πιστοποιητικών μπορεί να ανανεωθεί από 10 στα 15 χρόνια. Για την ETF θα θέλαμε αυτή η περίοδος να περιοριστεί στα 10 χρόνια. Θέλουμε τα πιστοποιητικά να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτά. Από εμένα και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο, ο κύριος Ρόμπ Φαν Ρέιμ από την Εντίνα, εκπαιδευτικό δίκτυο των, ε, των σχολών ε, εκπαίδευσης για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Καλημέρα. Η Εντίνα εκπροσωπεί τις σχολές εσωτερικής ναυσιπλοείας στην Ευρώπη. Η Εντίνα είναι πάρα πολύ ε, σύμφωνη με την πρόταση αυτή, την είχαμε υποστηρίξει από την αρχή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πρόταση. Μια πρόταση η οποία πηγαίνει σε ένα σύστημα το οποίο φεύγει από την εμπειρία μόνο και πηγαίνει και στις δεξιότητες. Αλλά θα εξακολουθεί βεβαίω και η εμπειρία ε, να παίζει ρόλο και, και να υπάρχουν και οι άλλε δοκιμασίες και τεστ και έτσι θα έχουμε υπεύθυνου ανθρώπου στην εσωτερική ναυσιπλοή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κλάδο τον δικό μας, ειδικά όσον αφορά την κατάρτιση. Θεωρούμε επίσης πάρα πολύ ε, σωστό το ότι αν έχουμε μία ε, οδηγία θα είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταφραστεί σε όλους ε, στο πρόγραμμα το διδακτικό στην ύλη και θα είμαστε σίγουροι ότι όπου και αν εκπαιδεύεται κανείς στην Ευρώπη θα είναι ικανός. Υπ' αυτήν την έννοια δεν αντιλαμβανόμαστε πλήρως το ότι σε κάποια σημεία αυτής της οδηγίας γίνεται λόγος για την δυνατότητα γραπτής εξέτασης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο σε συνδυασμό με τεστ γραπτής εξέτασης με τεστ γνώσεων και βεβαίως τεστ των ικανοτήτων. Υπάρχει λοιπόν κάποιο περιθώριο βελτίωσης ε, των προτάσεων της οδηγίας. Η οδηγία λέει πως περιορίζεται μόνο στο πλήρωμα του καταστρώματος και όχι της μηχανής. Μόνο που... Κοιτάξτε, εδώ πέρα, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη, δεν υπάρχει αυτός ο αυστηρός διαχωρισμός ε, κουβέρτα και μηχανή. Ε, το πλήρωμα τα κάνει όλα. Είναι και στην ε, γέφυρα και στη μηχανή. Οπότε θεωρούμε πως ο ναύτης θα πρέπει να εκπαιδεύεται και σε όλες τις πτυχές, όχι μόνο στα τρία πράγματα τα οποία αναφέρονται εδώ. Θα θέλαμε λοιπόν και για τους 7 τομείς ε, που υπάρχουν στον κλάδο μας να υπάρχουν αυτές οι διατάξεις. Για να μην τώρα έχουμε το φαινόμενο να υπάρξει διαφορετική μετάφραση σε κάθε κράτος μέλος ε, και να μην μπορούμε να βασιστούμε στην ομοιομορφία καλό θα είναι να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο θα εγγυάται την ποιότητα ακριβώς. Έτσι ώστε ε, και οι σχολές να έχουν ένα κοινό μέτρο αξιολόγησης. Κατόπιν, υγεία, όπως είπαμε, ε, αγγίζει και κάποια θέματα αρμοδιοτήτων. Και λέτε μάλιστα πως θα υπάρχουν και κάποια τεστ για την ικανότητα του ναυτικού να, δείξει, να επιδείξει ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε κυρίως για ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από άλλα επαγγέλματα και λέμε ότι θα πρέπει να έχουν πρώτα μία πενταετή εμπειρία για να μπορούν πρώτα απ' όλα να δηλώσουν ενδιαφέρον για αυτή τη δουλειά ή να γνωρίζουν ε, μία διαδρομή Βεβαίω υπάρχει το θέμα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε πάρα πολύ μικρές διαδρομές ε, ε, χωρίς να σημαίνει πως έχουν οπωσδήποτε πενταετή ε, εμπειρία. Και δεν βλέπω το πρόβλημα κάποιος ο οποίος είναι 21 ετών να πρέπει να, και έχει μόλις τελειώσει κάποια, κάποια σχολή, να του πούμε πήγαινε να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία και ποια εργασιακή εμπειρία. Αυτά. Ευχαριστώ. Επόμενος και τελευταίος ε, ένας μιλητής από την Επιτροπή του Ρήνου. Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα ως Κεντρική Επιτροπή για την Αυσιπλοεία στο Ρήνο να σας ε, μιλήσουμε για το σχέδιο οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα στην εσωτερική ναυσιπολη... ναυσιπλοεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η αμοιβαία αναγνώριση αρμοδιοτήτων. Έχει μακρά ε, παράδοση. Το 1922 η ΣΥΣΥ ενάρχθη στην πρώτη συμφωνία με τα κράτη-μέλη ε, σε όλη τη λεκάνη του, του Ρήνου ε, ξεκινώντας από τη Βασιλεία. Υπήρξε λοιπόν αμοιβαία αναγνώριση. Από τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε και έφτασε σε αυτή την κοινή πιστοποίηση Αναγνώρισε όλα τα επαγγελματικά προσόντα και τα πιστοποιητικά, την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων με την οδηγία 96 50 και αυτό στην, όσον αφορά την εσωτερική ναυσιπλοεία και αυτό αφορά και την ασφάλεια και ειδικότερα την ασφάλεια των επιβατών. Αυτά τα θέματα ανέπτυξε η CCNR σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις διαβουλεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής αναπτύχθηκαν περισσότερες, μάλλον προσθέθηκαν περισσότερες αρμοδιότητες στα παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη λεκάνη του Ρήνου. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναπτύξουμε πρότυπα για την λεπτομερή περιγραφή αρμοδιοτήτων, κάτι που προβλέπεται από την ίδια την οδηγία. Έχουμε ορισμένα ζητήματα εδώ σε σχέση με την πρώτη ε, εισαγωγή των ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων ε, για τους επωνομαζόμενους boatmen. Εδώ θα θέλαμε να δούμε ε, και να συνεργαστούμε με τους κοινωνικούς εταίρους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να συνεργαστούμε και να φτάσουμε σε κοινά πρότυπα και σε ε, ε, λειτουργικό επίπεδο και σε επίπεδο διαχείρισης. Χαιρόμαστε λοιπόν γιατί μπορούμε να συνεργαστούμε με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό αφορά και τις ειδικέ αδειοδοτήσεις, στις οποίες αναφέρθηκε ο εισηγητής. Θα πρέπει να δούμε περισσότερα ζητήματα, να τα δει δηλαδή ο νομοθέτης και όπως είπε και η συγγήτρια, θα πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία με την Επιτροπή αργότερα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτές τις προδιαγραφές. Βεβαίως, ε, είδαμε ότι δεν θα πρέπει να μειωθούν οι προδιαγραφές, δεν είναι η πρόθεση των κρατών μελών και του τομέα. Είναι κοινή αυτή η θέση και ακούσαμε και την ETF που ανέφερε το γεγονός ότι αυτή η οδηγία θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ποιότητας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι θα συνεισφέρουν σε αυτές τις ε, προδιαγραφές, αυτά τα κοινά πρότυπα. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πλαίσιο καθώς και οι χρονικές προθεσμίες χρειάζονται κοινέ προσπάθειες και χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων που προέρχονται από τα εκπαιδευτικά κέντρα για να δούμε πώς αναπτύσσονται και τα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα βασιζόμενο στα επαγγελματικά προσόντα. Χαιρόμαστε που είμαστε και εμείς μέρος αυτής της προσπάθειας και θα βοηθήσουμε το Κοινοβούλιο εάν χρειαστεί την υποστήριξή μας και χαιρόμαστε που διανοίγουμε αυτή τη δυνατότητα σήμερα. Ευχαριστώ που τηρήσατε και τα χρονικά όρια. Να ακούσουμε τον Κύριο Φαντερκάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος ο Ρενό Μιζελιέ δυστυχώς έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Είναι σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ για το θέμα αυτό και μου ζήτησε σήμερα να μεταφέρω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελε να συγχαρεί την Κομισιόν και να πει πως είναι θετική η πρόταση αυτή. Ακούσαμε και τους ε, ειδικού ε, και ξέρετε πως ε, το θέμα αυτό μας απασχολεί εδώ και δεκαετίες για να γίνει πιο επαγγελματικός ο κλάδος με εκπαιδευμένο προσωπικό και θέλουμε να έχουν την δυνατότητα να μπορούν ευκολότερα να δουλεύουν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν να δούμε σοβαρά την έλλειψη πληρωμάτων. Μιλάμε για modal shift, θέλουμε οι μεταφορές να μετατοπιστούν και προς τα ποτάμια και η έλλειψη πληρωμάτων είναι ένα θέμα και συνεισφέρει νομίζω αυτή η πρόταση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Κομισιόν τώρα μιλάει για μια εκπαίδευση με βάση τις ε, δεξιότητες. Είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε, αλλά βεβαίως έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Τις εξής πέντε. Πρώτον, το θέμα των ορισμών και συγκεκριμένα των εσωτερική της εσωτερικής ναυσιπλογίας και των πλεύσιμων ποταμών. Στο παράρτημα ορίζονται ε, διαφορετικές ζώνες εσωτερικής ναυσιπλογίας. Αλλά δεν τα βλέπουμε αυτά μετά στην πρόταση της οδηγίας. Την... Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. πέρα από το βαθμό εκπαίδευσης χρειάζεται για κάθε μέλος του πληρώματος μια πιστοποίηση. Το ερώτημα λοιπόν είναι πως είναι δυνατόν για κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους να μπει στο βιβλίο του καταστρώματος ότι είναι αυτά τα άτομα πλήρωμα με αυτές τις δεξιότητες και αυτά τα προσόντα. Τρίτο, ο χρόνος ε, στον εξομοιωτή, αν μετράει και αυτό το χρόνο εκπαίδευσης. Θέμα εκπαίδευσης, δηλαδή αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο είπε ο εκπρόσωπος των σχολών για τις γραπτές εξετάσεις, αλλά σκεφτόμαστε αν ε, θα μπορούσε να προσμετρήσει και ο χρόνος στον εξομοιωτή. Μετά έχουμε την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων, κάτι το εξαιρετικό ως μέσο, αλλά βεβαίω ε, υπάρχει και το ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και τέλος, υπάρχουν οι εποχιακοί εργαζόμενοι. Αποκλείονται αυτοί από το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ich danke auch. Und die nächste ist Anna Claudia. Ευχαριστώ, Άννα Κλαουδία Ταρπατέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο την εισηγήτρια καθώς και τους εμπειρογνώμονες για τις πληροφορίες που μας έδωσαν που είναι πολύ χρήσιμες. Σίγουρα η εσωτερική ναυσιπλοεία είναι ένας τρόπος οικονομικής ανάπτυξης όλων των παράκτιων περιοχών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε και με ένα βιώσιμο μέσο μεταφορών. Μιλάμε λοιπόν για δημιουργία ενός κοινού πλαισίου κανονισμών που να είναι ενιαίο. Γι' αυτό θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ τις προσπάθειες της Επιτροπής να ορίσει ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας μέσα στα πλαίσια της αμοιβαία αναγνώρισης αυτών των εγγράφων. Θα πρέπει να φτάσουμε και εδώ σε μία ενιαία αγορά και να μπορέσουμε να εξελίξουμε και τα επαγγέλματα και τις σταδιοδρομίες αυτού του τομέα. Θεωρώ λοιπόν ότι η εναρμόνιση της νομοθεσίας είναι σκόπιμη για όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν όμως δύο ερωτήματα, δύο ζητήματα που μας απασχολούν. Αφορούν τους, ε, τομείς που μπορεί να ενέχουν κινδύνους στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Δηλαδή δεν έχουμε ορίσει αυτές τις ζώνες κινδύνου ή επικινδυνότητας και γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε αυτά τα κριτήρια από κοινού. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι και η ε, συντήρηση αυτών των οδών από τις ε, αρμόδιες υπηρεσίες και γι' αυτό θα πρέπει ε, αυτές οι αρμοδιότητες να ενταχθούν στο άρθρο 8. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι επικίνδυνες ε, ζώνες ενέχουν και ένα επιπρόσθετο κόστος για τα κράτη-μέλη. Η δεύτερη πτυχή σχετίζεται με την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών αυτών επαγγελματικών προσόντων από την Επιτροπή του Ρήνου. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε έναν πιο απλό τρόπο αμοιβαία αναγνώρισης. Δηλαδή θα πρέπει να αρθούν τα γραφειοκρατικά προσκόμματα, να αναγνωρίζονται τα προσόντα και να μπορεί ελεύθερα να μετακινείται το εργατικό αυτό δυναμικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα μια πολύ καλή συνεργασία με την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε. Voorzitter, goedemorgen. κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση εδώ. Και βεβαίω η μεγάλη διαφορά είναι αυτό ακριβώς η πείρα και οι δεξιότητες. Και βεβαίω το θέμα των δεξιοτήτων είναι το πώς θα εφαρμοστούν στον τομέα της εκπαίδευσης. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάτι διαφορετικό, τον Ρήνο και την Επιτροπή του Ρήνου. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο μου ερώτημα αφορά το άρθρο 6, στο άρθρο 6 της πρότασης. Γίνεται λόγος για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που μπορούν να τεθούν ε, σε ναυτικούς ε, και καπετάνιους, ειδικά για νερά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αμέσως προκύπτει το ερώτημα τι γίνεται με τον Ρήνο. Ειδικά καθώς το Ρήνο πρέπει να γνωρίζει κανείς τη διαδρομή της ε, Κίτης. Και πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη διαδρομή όπως είπα. Και βλέπουμε στο άρθρο 6 πως τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ειδικέ άδειες ε, για κάτι τέτοιο ε, μπορούν να κάνουν αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα μη κράτος μέλος, η Ελβετία συγκεκριμένα. Τι γίνεται λοιπόν ε, με, την, με τις άδειες αυτές. Πρέπει να υπάρξει κάποια συμβουλή νομίζω. και δεν υπάρχει κάποια επιλογή ακριβώς στο άρθρο 6 για την ξεχωριστή ζώνη του Ρήνου. Δεύτερο ερώτημα. Οι εξομοιωτές. Κάπου παρακάτω στην πρόταση μιλάμε για τους ε, εξομοιωτές ε, άρθρο 19 σημείο 2 που λέει πως η Κομισιόν έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει την εκπαίδευση εξομοιωτές. Καλό είναι βεβαίως ε, να δουλεύουμε με εξομοιωτές, ναι βεβαίως, αλλά η εξομοίωση πάλι είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να ακούσω τι άποψη έχει γι' αυτό η ε, Επιτροπή του Ρήνου. Αυτές τις ε, δύο ερωτήσεις για τον ε, Ρήνο και μια άλλη ακόμα ερώτηση. Έχοντας ακούσει τον εκπρόσωπο του ETF, έχουμε το άρθρο 5, άρθρο 10, με συγχωρείτε, 5, όπου μιλάμε για μια δεκαετή περίοδο. Θα ήθελα να μάθω η Κομισιόν πώς το βρήκε αυτό τον αριθμό. Εντάξει, ωραία, ακούγεται 10 χρόνια Ποια είναι η λογική πίσω από αυτό. Αυτά. Σας ευχαριστώ και αναμένω βέβαια και τη συνεργασία με τους άλλους και ηγητές και την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Keith Taylor, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίζουμε αυτή την προτινόμενη οδηγία γιατί θα αντικαταστήσει μία ε, πολυσχηδή σειρά περιφερειακών απαιτήσεων με απλούστερες. Πρόκειται λοιπόν για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης. Άκουσα τι είπαν οι εμπειρογνώμονες και δεν νομίζω ότι είναι παρόντες όλοι οι τομείς εδώ γι' αυτό. Θα ήθελα να ε, μιλήσουμε περισσότερο για την εσωτερική ναυσιπλοεία της Ευρώπης γενικότερα. Τι πιστεύουν οι εμπειρογνώμονες για τις ελάχιστες προδιαγραφές κατάρτισης στα πλαίσια της ασφάλειας των επιβατών κατά την ναυσιπλοΐα; γιατί είχα, ε, έχω συντάξει μάλλον και μία ε, πρόταση σε σχέση με την οδηγία για την εσωτερική ναυσιπλοεία και την ασφάλεια των επιβατών. Τι πιστεύετε ιδιαίτερα για τους ανθρώπους με αναπηρίες και με περιορισμένη κινητικότητα. Θεωρείτε ότι η μελέτη αντικτύπου της Επιτροπής αρκεί και φτάνει σε συμπεράσματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες μας. Τώρα, ως προς την Επιτροπή, πώς θα αποφύγουμε αυτή τη διτή ρύθμιση για το μέλλον, για να μην υπάρχουν επικαλύψεις στην εργασία μας και διοικητικός φόρτος προς τα κράτη-μέλη. Τι σκέπτεστε για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για την εσωτερική πλωτή ε, για την εσωτερική ναυσύπλοεία και για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Όπως αναφέρει και η CCNR, η Επιτροπή για την Ναυσύπλοεία του Ρήνου, τι σκέφτεστε ως προς τα δεδομένα του κοινωνικού ε, διαλόγου σε σχέση με το ημερολόγιο πλεύσης και τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε ηλεκτρονικά, έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε μία συνολική εικόνα για τα τεκτενόμενα. Ελπίζω να φτάσουμε σε κάτι πολύ θετικό από την οδηγία αυτή, όπως θα εξελιχθεί. Ιζαμπέλα Ντεμόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους εμπειρογνώμονες που μας μίλησαν για το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας. Καταρχήν, για την κινητικότητα των εργαζομένων θα πρέπει να κινηθούμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση εποπτείας και σταθερότητας ως προς τις θέσεις εργασίας για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ως προς το περιεχόμενο τώρα, μιλάμε για μία οδηγία και αφήνουμε περιθώρια στα κράτη-μέλη να κινηθούν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους και το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο στο ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει υπερβολική ευελιξία. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, στο σύστημα εξαιρέσεων δεν θα πρέπει να φτάσουμε σε νομική ανασφάλεια. Ως προς τις ερωτήσεις, η μία φορά τις εξαιρέσεις, την εξαίρεση από την αξιολόγηση. Δεν θα ήταν σκόπιμο να μιλήσουμε για την ε, πείρα ναυσιπλοείας παρά για επαγγελματική πείρα γενικότερα. Και στον τομέα της κατάρτισης, στο άρθρο 17 βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, κοινοποιούν τα προγράμματα πώς θα μπορούσαμε να έχουμε εγγυήσει και ποιοτικά αποτελέσματα για να υπάρχει ένα ομοιογενές πλαίσιο λειτουργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε. Ετέθησαν κάποια ερωτήματα, όχι προς την εισηγήτρια βέβαια, αλλά προς τους παρεμβαίνοντες. Αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε. Να ακούσουμε την ε, κυρία Χακστάινα πρώτα, με τη σειρά. Ευχαριστώ για όλη σας την στήριξη και για τα ερωτήματά σας. Κατανοώ ότι από τη μία υποστηρίζετε την προσέγγιση, αλλά εκφράζετε κι εσείς κάποιες ανησυχίες. Νομίζω ότι πολλά από τα ερωτήματα ε, κυρίως απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά για τα ερωτήματα, για να ξεκινήσω από το τέλος, ο κύριος Τέιλορ έθεσε κάποια ερωτήματα για την επιβετικά σκάφη και τα πρότυπα για τις επίγουσες καταστάσεις και τι γίνεται με την κινητικότητα. Βεβαίω, στον ε, τομέα αυτό ήδη έχουμε πολύ υψηλό πρότυπο ασφάλειας, αυστηρό. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε υψηλό επιπέδου ασφαλεία και θεωρούμε ότι τα πρότυπα που υπάρχουν είναι επαρκή για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες. Σε σχέση τώρα με το διοικητικό άχθος, είναι όντως και αυτό ένα θέμα που θέλαμε και εμείς να το δούμε. Κάτι άλλο που είπανε κάποιοι ευρωβουλευτές ήταν το θέμα του κινδύνου και τι γίνεται με τις εξαιρέσεις. Όντως για εμάς ως ε, κλάδο ε, είναι σημαντικό να τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες και αντίθετα με τα όσα είπαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό για μας να υπάρχουν κάποιοι, α, ε, παρά, κάποιοι τομείς όπου να μπορεί να υπάρχει ακόμη πιο υψηλή ασφάλεια. Ας πούμε για περιπτώσεις ε, ατυχημάτων που μπορεί να γίνουν. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απαραίτητες ε, δικλείδε ασφαλείας. Το πρότυπο που έχει η CCNR πρέπει να διατηρηθεί για την ασφάλεια και βεβαίως να εμπλουτιστεί. Και αυτό σίγουρα θα οδηγήσει σε μείωση της γραφειοκρατίας. Τώρα για τους εξομοιωτές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από τη μια την ε, εμπειρία αυτή, αυτή τη, αυτής της μοντέρνας τεχνολογίας, αλλά αυτή πρέπει να συμβαδίζει και με την πρακτική κατάρτιση, εκπαίδευση ε, επί των σκαφών. Και πρέπει εδώ να βρούμε μια λύση έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε στο υψηλό πρότυπο ασφαλείας. Ε, νομίζω ότι έχω απαντήσει στα ερωτήματα. Νομίζω. Αυτά, πρόεδρε από μένα, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Μίριαμ Σεφάρ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι με όλα τα σχόλια και τα δεδομένα και το feedback Η θέση μας είναι πιο διευρυμένη σε σχέση με αυτά που παρουσιάσαμε και στην πρώτη μας ε, εισήγηση, αλλά χαίρομαι γιατί μιλήσατε για ψηφιακούς ταχογράφους. Είναι κάτι το οποίο είχαμε ζητήσει και εμείς και θα θέλαμε να τεθεί σε εφαρμογή με όλες, ε, με όλα τα άλλα μέτρα αν θέλουμε η βιομηχανία να είναι πιο βιώσιμη, λίγο πιο βιώσιμη έτσι ώστε να ε, εποπτεύουμε τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης. Δεν πρόκειται για έναν τόπο εργασίας, αλλά και τόπο διαμονής για τους εργαζόμενους για μακρά χρονικά διαστήματα. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς και ποιους ορίζουμε και οριοθετούμε ε, αυτή την οδηγία. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να καλύψουμε όλες τις εργασίες, δηλαδή και το προσωπικό που δεν ασχολείται άμεσα με την αυσιπλοεία. Πολλές φορές μιλήσαμε για εποχική εργασία και πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι έχουν συμβόλαια εννέα μηνών, αλλά εργάζονται πολύ περισσότερες ε, ώρες σε εννέα μήνες από ότι εμείς σε δώδεκα. Είναι λοιπόν πλήρης η απασχόληση και θα πρέπει να ε, αμείβεται σωστά να υπάρχει αξιοπρέπεια σε αυτή την εργασία και να μην βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι σε μια κατάσταση πλήρους ε, ευαλωτότητας με πολύ χαμηλότερους ε, μισθούς. Ως προς τους προσωμιωτές αναφέρθηκαν ήδη θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε και στα πλαίσια της εσωτερικής ναυσιπλοείας με αυτά τα μέσα γιατί είναι ένας τρόπος ε, διδασκαλίας, ε, ε, διδαχής δεξιοτήτων. Εάν οι άνθρωποι εκπαιδευόμενοι έχουν σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης, αυτά τα μέσα θα αποδώσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουν ουσιαστική πείρα ναυσιπλοείας, αλλά οι προσωμιωτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Ε, ο συνάδελφός μου από την Εντίνα μίλησε και για τις αρμοδιότητες δυνάμει αυτής της οδηγίας. Θα θέλαμε και οι επτά οριζόμενες ε, ε, δεσμεύσεις να, να ενταχθούν εδώ και όχι μόνο οι τρεις που αναφέρονται στο άρθρο 3. Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, αλλά μπορείτε να τις δείτε στο γραπτό μας που έχουμε υποβάλει. Mm. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ σε κάποιες ερωτήσεις που σημείωσα. Να εκπαιδευτούν όλα τα μέλη του πληρώματος ή όχι. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή η οδηγία αφορά το πλήρωμα των καπετάνιων και τους ε, ε, ναύτες. Σε αυτούς περιορίζεται. Αυτό το οποίο ξέχασα ε, είναι ότι μιλάμε και για την ασφάλεια, την ασφάλεια των ανθρώπων που δουλεύουν στον ε, κλάδο και την ασφάλεια γενικά της ναυσιπλογίας. Οπότε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως κάποιος ο οποίος ε, δεν έχει καμία γνώση του θέματος μπορεί να ανέβει σε μια τέτοια λάτζα σε ένα τέτοιο πλοίο. Γιατί βλέπουμε ότι για έναν απλό ναύτη ε, αρμενιστή δεν υπάρχει καμία απολύτως απέτηση. Ε, υπάρχει για τον οποιονδήποτε είναι πλήρωμα σε πλοίο η απέτηση να γνωρίζει τα ελάχιστα περί κινδύνου και ασφάλειας. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει μια βασική εκπαίδευση ασφάλειας όσον αφορά τώρα τους ε, εξομοιωτές. Ναι. Έχουμε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο στην Εντίνα, όπως το λέμε. Δηλαδή, τι, πώς το λέμε εμείς, λέμε ακούω και ξεχνάω, βλέπω και καταλαβαίνω κάνω και το μαθαίνω. Δηλαδή χρησιμοποιούμε εκπαιδευτικά πλοία για να κάνει ο κόσμος πρακτική και εξομοιωτές ε, και χρησιμοποιούμε εξομοιωτές ε, και για τις ε, μανούβρες και για την ευσυπλογία αλλά και για τις άλλες λειτουργίες του πλοίου και είναι ελκυστικό αυτό για τους εκπαιδευόμενους και μαθαίνουν έτσι δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε ένα σχετικό σχέδιο ήδη από πολλές δεκαετίες. Είχαμε λοιπόν ένα έγγραφο το οποίο αναπτύξαμε για τον εξομοιωτή γέφυρας και με βάση αυτό ε, έχουμε και άλλες προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές ε, που θα πρέπει να πληρούν ε, οι εξομοιωτές, δηλαδή να εξομοιώνουν επαρκώς την πραγματικότητα για να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για εκπαίδευση αλλά και για αξιολόγηση του εάν κάποιος κατέχει τις δεξιότητες που πρέπει. Λοιπόν, όσον αφορά το πλήρωμα επιβατικών πλοίων, πράγματι παίζει ε, ένα ε, μάλλον στις περιπτώσεις που παίζει ένα ρόλο αυτό για το πλήρωμα θα πρέπει να υπάρχει βεβαίως μια σχετική πιστοποίηση. Στην περίπτωση που δεν τους αφορά δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Ε, το προφανές δηλαδή να μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε περίπτωση ανάγκης. Λοιπόν, Στις υφιστάμενες ε, λοιπόν δεξιότητες όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή και σε επιχειρησιακό επίπεδο και στην εκπαίδευση ε, προβλέπεται και νομίζω πως η οδηγία έχει κάνει εδώ πέρα την επιλογή να έχει ένα διαφορετικό ξεχωριστό τμήμα. Αυτή είναι η πρόταση. Η αμοιβή αναγνώριση τώρα. μεταξύ των κρατών που βρέχονται από τον τα οποία διατρέχει ο Ρήνος. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το οποίο λέμε τι γνώσει ε, συγκεκριμένων τμήματων της διαδρομής, αλλά υπάρχει και η βασική γνώση που θα πρέπει ε, να την ε, κατέχουν ε, όλοι για να μπορούν να ανταποκριθούν στις γενικότερες απαιτήσεις της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Μετά. Για να δω. Ναι, για το ημερολόγιο καταστρώματος. Ε, ξέρετε πως πάμε και στα ναυτικά φυλάδια και στο ημερολόγιο καταστρώματος σε μια ψηφιοποίηση και ψηφιοποίηση και τυποποίηση έτσι ώστε και τα ναυτικά φυλάδια και τα ημερολόγια καταστρώματος να είναι ηλεκτρονικά. για να υπάρχει και ένα άλλωστε ναυτικό φυλάδι να μην έχει κανείς ε, την υπηρεσία του καταγεγραμμένη σε πέντε διαφορετικά πλοία. Μετά, η ναυσεπλοεία. Κοιτάξτε, ε, συγκεκριμένα δηλαδή η ναυτιλία κατεύθυνση, όπως τη λέμε θα πρέπει πράγματι να αποδείξει κανείς με τεστ ότι είναι ικανός ή να αποδείξει εμπειρία από άλλους ε, κλάδους, από άλλους κλάδους της ναυτιλίας πάντα, έτσι. Έτσι αποδεικνύεται η ικανότητα, αλλά το μέτρο είναι αν κάποιος είναι ικανός ή όχι. Είναι ναι ή όχι. Αυτά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Uh, Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, το βασικό θέμα είναι η, διπλή εργασία, η ΣΕΣΝΗ που κατάρτισε τα πρότυπα στην εσωτερική ναυσιπλοεία, η ΣΕΣΝΗ, έχει σαν στόχο να αποφύγει την ε, ε, διπλή αυτή εργασία. και τη στιγμή που όλοι τηρούμε τις ίδιες προδιαγραφές, τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές, δεν νομίζω ότι θα έχουμε επιπρόσθετη γραφειοκρατία. Θέλουμε να φτάσουμε σε καλά αποτελέσματα και να μην υπάρχει επικάλυψη εργασίας. Αυτό θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί. Υπάρχει περιθώριο ε, εργασίας, μιλάμε για τους ε, προσωμιωτές, την ενδεχόμενη ε, χρήση τους, που θα υπόκεινται βεβαίως σε κανόνες και βεβαίως και η έγκρισή τους, γιατί θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια είναι τα ευεργετήματα της χρήσης των προσωμιωτών. Για να δούμε κατά πώς υπάρχει αντιστοιχία με συγκεκριμένες ε, δεξιότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι και διμερώς θα μπορέσουμε να δούμε ζητήματα τα οποία δεν μας απασχόλησαν εδώ. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Γιάν Σίμονς από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τον εισηγητή. Eh, eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ε, εισηγητής ε, για αυτό το θέμα. Ήδη πριν από αρκετά χρόνια είχαμε στις Ναϊάδες τον σχετικό κανονισμό ασχοληθεί με το θέμα και είχαμε έρθει και σε συνεννόηση με την Επιτροχή του Ρήνου. Χαίρομαι για την έντονη ενασχόληση με το ζήτημα και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Κομισιόν σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη Ε, η οποία ακόμα βέβαια δεν έχει καταλήξει επισήμως ε, στο πλαίσιο της ε, ΣΕΣΝΗ. Λοιπόν, δεν θέλω να επαναλάβω τώρα τα όσα είπαν οι ειδικοί για τις προδιαγραφές ασφαλείας, τη, μετα... τη μετάβαση από την εμπειρία στις δεξιότητες ναι. Είμαι όμως ε, υποχρεωμένος να αναπτύξω κάποιες σκέψεις ε, που έχουμε ε, για να τις έχετε κι εσείς υπόψη σας. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα το pacta sunt servanda. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πως πουθενά δεν γίνεται λόγος για την ε, συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με το CCR ως ε, διεθνή ως διεθνής οργανισμός ο οποίος έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τον Ρήνο. Ο κύριος Φαντάλεν μόλις βεβαίως εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και θα ήθελα να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, γιατί η αφετηρία μας εδώ πέρα είναι να υπάρχει μια αναγνώριση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να εξηγούμε μετά ποιες είναι οι εκτελεστικές ε, αρμοδιότητες. Υπάρχει βεβαίως και η πράξη του Μανχάιμ με το άρθρο 23, αλλά υπάρχει και το πρωτόκολλο 7 και το πρωτόκολλο 10 με τις σχετικές εξηγήσεις στο σημείο 1 και 2, το οποίο ξεκαθαρίζει τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής του Ρήνου για τον Ρήνο. Αν δει κανείς μετά το άρθρο 351 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, το οποίο αναφέρεται στην πράξη του Μανχάιμ, η οποία σας υπενθυμίζω είναι 200 ετών η συνθήκη. Ε, αναφέρεται λοιπόν πως η, άλλη συνθήκη προηγείται και αν σκεφτείτε πως είναι συμβαλόμενο μέρος ε, και η Ελβετία στην πράξη του Μανχάιμ, αλλά δεν είναι κράτος μέλος ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μόνο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε δυσκολίες στην εσωτερική ναυσιπλοεία, ειδικά αν διακατεχόμεθα από ευρωπαϊκό πνεύμα. Η λύση λοιπόν είναι απλούστατα. Οι άλλες ε, τέσσερις επιτροπές που έχουν αποκλειστικές αρμοδιότητες να περιληφθούν ε, στον κανονισμό και να πούμε ότι μπορούν να περιγράψουν τους συγκεκριμένους ε, κινδύνους, ότι μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα, να καθορίζουν τους κανόνες τους ανεξάρτητα και οπωσδήποτε σύμφωνα με την ε, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς είμαστε διατεθειμένοι εδώ πέρα να παίξουμε έναν ρόλο καταλήτη. Ευχαριστώ. Τώρα, έγιναν πολλές ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Το λόγο έχει ο κύριος Θεολογίτης. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning, ladies. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα με την μεγάλη υποστήριξη από όλες τις πλευρές για την ε, πρωτοβουλία μας. Αυτό δείχνει ότι στην ανακοίνωση Ναϊάδες του 2013 για τα ποιοτικά πρότυπα στην αυσιπλοεία αντικατοπτρίζεται σε αυτή την πρόταση. Επίσης, ε, κατά τη δημιουργία αυτής της πρότασης, ο κύριος ε, Χάγκεν και η Κριστέλ Ρουσό ε, συνεργάστηκαν με τον τομέα, τα κράτη-μέλη, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ούτω καθεξής. Και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα. Δεν λέμε ότι είναι τέλειο αυτό το πλαίσιο εργασίας. Μπορεί να βελτιωθεί. Θα ακούσουμε και το Συμβούλιο και θα εισαχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση η οποία θα εμπλουτίσει την πρόταση ποιοτικά. Είναι κάτι που προσφέρει η Επιτροπή στον τομέα αυτό για να δούμε ε, κατά πόσο τα πληρώματα είναι ακόμα ανεπαρκή, λαμβάνοντας υπόψη τη γύρανση του πληθυσμού και του, της μέσης ηλικία των πληρωμάτων και τις διαφορές που είχαμε μεταξύ της Επιτροπής του Ρήνου και των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων της Ευρωπαϊκής ε, Πιστοποίησης. Δεν έχει σημασία σε ποιον έγκυται, πού βρίσκεται η αρμοδιότητα επακριβώς και ποιος είναι υπέτειος για τα λάθη. Αλλά συμφωνήσαμε με τις, την Κεντρική Επιτροπή του Ρήνου να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο αυτής της οδηγίας, δηλαδή την κινητικότητα του, των εργαζομένων και η προσέλκυση νέων στο επάγγελμα. Για να απαντήσω τώρα σε μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν, φυσικά υπάρχουν περισσότερες δεξιότητες ε, που αφορούν το μηχανικό εξοπλισμό και άλλα ζητήματα που ασκούνται από το πλήρωμα, αλλά θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα, τις απαραίτητες δεξιότητες από αυτές που ασκούνται. Γι' αυτό έχουμε ένα απλό σύστημα μικρών περιορισμένων κατηγοριών που θα πρέπει να κατέχουν ένα εύρους δεξιοτήτων, όπως περιγράφεται στα παραρτήματα. Και εδώ έχουμε και κοινή συνεργασία με τις Επιτροπές ε, Εσωτερικής Ναυσιπλοείας και με τη ΣΕΣΝΗ που ε, προσδιορίζει τα πρότυπα και τις ε, προαπαιτήσεις που θα μας αναφέρετε εσείς ως ε, νομοθέτες από κοινού. Ως προς τα πρότυπα ασφαλείας, οι εμπειρογνώμονες είναι εκείνοι οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μας για να φτάσουμε σε αυτή την πρόταση. Τώρα έχουμε ένα σύστημα που βασίζεται στις συγκεκριμένες αρμοδιότητες έτσι ώστε να υπάρχει υψηλότερο επίπεδο προδιαγραφών ασφαλείας και στο Ρήνο. Δεν λέμε ποιο είναι καλύτερο. Είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ακόμα υψηλότερα τον πύχη και αυτό ικανοποιεί τον τομέα τους πλειοκτήτες και το περιβάλλον μας. Ως προς τους εξομοιωτές, που είναι ένα ζήτημα που έχει περιγραφεί, χαιρόμαστε γιατί μιλήσατε για την ανάγκη εξυγχρονισμού. Οι εξομοιωτές είναι πολύ σημαντικοί για την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και ούτω καθεξής. Δεν ε, αντικαθιστούν όμως την πείρα εμπλό ε, σε σχέση με δύο-τρεις ώρες τον εξομοιωτή. Γι' αυτό αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε εξομοιωτές υψηλού επίπεδου. Μπορείτε να έχετε έναν εξομοιωτή και σε ένα κινητό σήμερα. Αυτό όμως δεν αρκεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια πραγματική εκπαίδευση σε εξομοιωτή, σε πραγματικό εξομοιωτή για την εσωτερική ε, ναυσιπλοεία. Μιλάμε λοιπόν και για την ε, εποχή της ψηφιοποίησης και όπως αναφέρεται και στο προήμιο αυτού του μέσου, ασχολούμαστε με τα ε, ηλεκτρονικά μητρώα και τα ηλεκτρονικά ημερολόγια καταστρώματος. Δηλαδή γίνονται τώρα δύο μελέτες, η μία ολοκληρώνεται που αφορά την ηλεκτρονική εσωτερική ναυσιπλοεία και θα προωθηθεί περαιτέρω για να φτάσουμε σε προτάσεις για να υπάρχει επαρκής ασφάλεια όταν εφαρμόζουμε αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα. Θα ήθελα να απαντήσω στην ε, Συνομοσπονδία Εργαζομένων Εσωτερικής ε, Ναυσιπλοείας. Όπως ξέρετε, μία νομοθετική πρόταση χρειάζεται μακρά προετοιμασία. Πρέπει να γίνουν ε, πολλές διαβουλεύσεις, να γίνει μια μελέτη αντικτύπου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά εργαζόμαστε έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ε, εργαζόμαστε με σπουδή. Ως προς τις ζώνες αυτές κινδύνου υπάρχουν φυσικά και ιδιαίτερα στα ποτάμια. Πρόκειται ε, για ζωντανούς οργανισμούς. Μπορούμε να έχουμε και παλήριες, παλιροϊκά κύματα, αλλαγές και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει διάκριση για το ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες, οι βασικές γνώσεις που σχετίζονται και με τη μορφολογία του ποταμού. Και γι' αυτό ορίσαμε κριτήρια που πρέπει να πληρούνται τη στιγμή που μία συγκεκριμένη ζώνη θεωρείται ζώνη κινδύνου. δεν θα θέλαμε να έχουμε πληθώρα ε, ζωνών, γιατί αυτό θα μπορούσε να μειώσει την κινητικότητα αυτών που θέλουν να ε, πλεύσουν σε αυτές τις περιοχές. Σε αυτά τα περάσματα. Τώρα, σε σχέση με τα πρόσωπα με περιορισμένη κινητικότητα, θα το λάβουμε υπόψη, θα εισαχθεί, θα ενταχθεί στον ορισμό των ε, προδιαγραφών για τις αρμοδιότητες και αυτό θα απασχολήσει και το ΣΕΣΝΗ έτσι ώστε να ενταχθούν αυτά τα πρόσωπα. και οι ανάγκες του στον κανονισμό. Τέλος, για την ανάγκη ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εσωτερικής Ναυσιπλοείας, όπως ξέρετε δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, ένας οργανισμός ε, χρειάζεται πολλή δουλειά πριν συσταθεί. Είχε γίνει τέτοια συζήτηση στο παρελθόν, το Κοινοβούλιο είχε σταθεί επικριτικό ακούσαμε και διαβάσαμε την έκθεσή σας κυρία Τέιλορ. Θα, θα λάβετε επίσημη απάντηση και θα ήταν σκόπιμο να παραμείνω εδώ και να μην επεκταθώ. Ελπίζω να απάντησα στα περισσότερα σχόλια και σε ερωτήσεις. Και τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επικοδομητική εργασία, όχι μόνο σήμερα, αλλά μέσα ε, στα πλαίσια συνεργασίας, της πολιετού συνεργασίας που είχαμε. Θα εισακουστείτε ως επιτοπλίστων υπάρχουν θέματα όχι μόνο τεχνικά αλλά και πολιτικής υφής. Γι' αυτό ε, επιθυμούμε το input από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τρίτες χώρες το θέμα αυτό. Οι συνάδελφοί μου και εγώ θα θέλαμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας επί του θέματος και ξέρουμε ότι και εσείς θέλετε να προχωρήσετε τάχιστα κάτι το οποίο θέλουμε και εμείς και το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. Και να ακούσουμε τώρα τελευταία πια την ε, εισηγήτρια, την κυρία Μάσινερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους ε, που ήταν παρόντες, ευχαριστώ που ακούσαμε την εμπειρογνωμοσύνη σας. Ε, νομίζω ότι ήταν πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ και τους σκιώδες ηγητές, όχι μόνο για τις προτάσεις τους που ακούσαμε σήμερα και ε, για τους καλεσμένους μας που μου πρότειναν να τους καλέσουμε σήμερα, αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που μας απασχολεί άλλους. Προφανώς υπάρχουν βεβαίως διαφορετικές απόψεις και διαφορετικά, διαφορετικές οπτυχές στα κράτη-μέλη. Ακούσαμε λοιπόν διάφορα διάφορα απόψει, μια στιγμή να πιω και μια γουλιά νερό. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια πολύ καλή έκθεση. Υπάρχουν πολλά θέματα να σκεφτούμε. Ακούσαμε και από του εμπειρογνώμονε ότι ουσιαστικά Τώρα η πρόκληση για μας και για μένα ως εισηγήτρια δεν είναι να ε, συγκεράσω όλες τις απόψεις μόνο των, κρατών, των ε, συναδέλφων, αλλά να δούμε τι είναι και σκόπιμο και για τον ε, κλάδο. Θέλουμε κινητικότητα, θέλουμε καλούς εργαζόμενους με γνώσεις. Ε, υπάρχουν διάφορα επίπεδα λοιπόν που πρέπει να συνδυαστούν. Υπάρχουν ε, κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, πρόσβαση σε άλλα κράτη-μέλη που έχουν πλωτές οδούς. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτό που είπε η ETF, ότι πρέπει όλοι να έχουν την ίδια εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το πού θα απασχοληθούν. Όλα αυτά λοιπόν είναι μεγάλη πρόκληση. Θέλουμε να έχουμε ευελιξία, δεν θέλουμε γραφειοκρατία, θέλουμε να μπορούμε να έχουμε ευκολότερη πέρασμα για τους ήδη εργαζόμενους εργαζόμενους στον κλάδο σε άλλα πόστα τι κάνουμε με τη μεταφορά επικίνδυνων ε, φορτίων, τι κάνουμε με τη μεταφορά επιβατών. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε κάτω από μια ευέλικτη και διαφανή προσέγγιση. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Ήδη ξέρω ότι θα υπάρξουν κάποια σημεία που πρέπει να τα συζητήσουμε ως ε, κοινοβούλιο και ίσως να χρειαστεί να αλλάξουμε λίγο τη θέση μας, αλλά είμαι αρκετά πεπισμένη ότι θα τα καταφέρουμε να φτιάξουμε μια καλή έκθεση. Είχα πει και, προ... Είχα πιο πριν ότι θέλω να έχουμε μέχρι το τέλο του έτους ολοκλήρωση της έκθεσης νομίζω ότι το Συμβούλιο ήδη είναι έτοιμο με την δική του τη γνωμοδότηση. Συνήθω δεν συμβαίνει αυτό. Το Κοινοβούλιο συνήθω είναι πιο γρήγορο από το Συμβούλιο. Τώρα δεν ξέρω, ίσω επειδή έχει να κάνει με νερό, ίσω επειδή έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη οδηγία, πήγε γρήγορα και το Συμβούλιο. Ε, και άκουσα μάλιστα ότι οι ε, κάτω χώρε πιέζουν πολύ για να υπάρξει μια κοινή ε, έκθεση, μια κοινή θέση από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της δικής τους Προεδρία. Ελπίζω και το Κοινοβούλιο να, ήθελα μόνο το Κοινοβούλιο να είναι εξίσου γρήγορο, αλλά δυστυχώ δεν μπορούσαμε να προλάβουμε όλες τις προθεσμίε κτλ. Οπότε καλό θα είναι να προχωρήσουμε από εδώ και μπρο γρήγορα, γιατί νομίζω ότι πραγματικά μιλούμε όλοι για το ίδιο πράγμα, για καλέ θέσει εργασία, με καλά προσόντα, με ασφάλεια και, με, μιλάμε για έναν κλάδο που πρέπει να αναπτυχθεί. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με όλες αυτές τις ε, ε λεπτομέρειες και να μην ε, ε, πάμε πιο γρήγορα από ό,τι είναι απαραίτητο ή από ό,τι μπορούμε. Χαίρομαι λοιπόν πολύ για την επόμενη συνάντηση που θα έχουμε με τους σκιώδεις ηγητές. Εγώ ήδη έχω κάνει πολλές συζητήσεις, φαντάζομαι και οι σκιώδεις μου επίσης και τις επόμενες ημέρες ε, θα έρθω σε επαφή με συναδέλφους, με εκπαιδευτικά κέντρα, θα δούμε τι γίνεται με τα εκπαιδευτικά σκάφη. Ε, και επίσης, ε, είναι κάτι που εμένα με απασχολεί ιδιαίτερα, θέλουμε να υπάρξουν θέσεις εργασίας για γυναίκες στον κλάδο αυτό, γιατί πάντα είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε άντρες, ε, να δουλεύουν στα σκάφη. Ε, πολλές φορές όμως ε, τα σκάφη αυτά είναι και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και οι γυναίκες δουλεύουν απλώς επειδή είναι παντρεμένες με τον καπετάνιο. Θα θέλαμε όμως να έχουμε και καλές θέσεις για γυναίκες. Στο μέλλον λοιπόν καλό θα ήταν ο κλάδος αυτός να μπορέσει να γίνει πιο ασφαλής και πιο ελκυστικός και να μπορεί να δραστηριοποιείται ο κόσμο σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης. Χαίρομαι λοιπόν και για την περαιτέρω συνεργασία μας. Ήδη υπάρχουν ε, πολλά πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε και βεβαίως προσβλέπω και στην ανταλλαγή απόψεων με τους ε, ε, εμπειρογνώμονες και στο μέλλον. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να δούμε τι θα καταφέρουμε να κάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ Γκέζινε Μάισνερ. Ήσουν πολύ ακριβής και ήσουν και εντός των χρονικών ορίων. Λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου θα περιμένουμε την έκθεσή σου και όσο πιο γρήγορα γίνεται όπως είπαμε, αλλά βεβαίως ε, να μην ε, κάνουμε και ε, τσαπατσούλικες δουλειές. Πάμε τώρα στην επόμενη, στο επόμενο σημείο, έλεγχος των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης μου θα μας ενημερώσουν για τα μέτρα, για τα, για τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου. Και όπως ξέρετε αυτά τα λειτουργικά τμήματα εδώ και χρόνια δεν έχουν εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη έτσι όπως τα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. εμείς από την Επιτροπή Τραν χρόνια συζητούμε το θέμα αυτά και το έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη να γίνει σωστή εφαρμογή. Θυμάμαι παλιότερου συναδέλφου, ε, μάλιστα ένα συνάδελφο που ήταν και συντονιστή και προσπαθούσε έντονα να προωθήσει αυτά τα ε, λειτουργικά ε, τμήματα του ενέργειου χώρου. Χρειαζόμαστε λοιπόν άμεσα πιο αποτελεσματική χρήση του ενέργειου χώρου μας, γιατί με την πιο αποτελεσματική χρήση μπορούμε να γλιτώσουμε και καύσιμα, να εξοικονομήσουμε χρόνο και να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων. Και στην ε, πολιτική, σε αυτό το τομέα έχουμε μια ε, ε, κατάσταση όπου μπορούν όλοι να κερδίσουν. Πρέπει να πάμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα ωφεληθούν μόνο οι επιβάτες που θα έχουν λιγότερες καθυστερήσεις και οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά και το περιβάλλον μας. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, χαίρομαι για την παρουσίαση που θα μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα λειτουργικά τμήματα του εναρίου χώρου, για το πώς αυτά μπορούν να εφαρμοστούν. Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Μαουρίτσιο Καστελέτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Ε, εντάχει θα θέλαμε να σας πούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτά τα λειτουργικά τμήματα και θα θέλαμε να σας πούμε ποιοι είναι οι άξονες ε, εργασίες, εργασίας σε σχέση με τον ε, ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Όπως ξέρετε, το σχέδιο απόδοσης η αποδοτικότητα είναι ένα κεντρικό μέσον, ένα βασικό μέσον, το οποίο ε, εισήχθη το 2009 μέσα στα πλαίσια του δεύτερου νομοθετικού πακέτου για τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ουρανό. Είναι ε, ένα μέσο που βοηθά τους ε, παρόχους υπηρεσιών, γιατί σήμερα λειτουργούν μονοπωλιακά και γι' αυτό δεν μπορούν να παρέχουν τις βέλτιστες υπηρεσίες στους τελικούς καταναλωτές και στην αγορά γενικότερα. Αυτό λοιπόν το σχέδιο απόδοσης είναι πολύ λεπτομερές και γι' αυτό προσπαθούμε να φτάσουμε σε, τόχους, σε στόχους απόδοσης για την ασφάλεια, περιβάλλον, ε, χωρητικότητα ή ικανότητα και αποδοτικότητα. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φτάσουν σε εθνικά σχέδια αποδοτικότητας με δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά αυτά τα λειτουργικά τμήματα για να ε, δείξουμε ότι αυτά τα ε, λειτουργικά τμήματα σχετίζονται με ευρωπαϊκούς ε, στόχους. Μετά την παράδοση των λειτουργικών τμήματων γίνεται αποτίμησή τους από την Κομισιόν με τον οργανισμό απόδοσης για την ε, συνολική αξιολόγηση και μετά εμείς εγκρίνουμε αυτά τα σχέδια απόδοσης ή όχι. Ανάλογα, αυτό γίνεται σε δύο φάσεις. Αρχικά μπορεί να ανακύψει αρνητική απόφαση της Επιτροπής. Εάν όμως αναθεωρηθεί από τα κράτη-μέλη ε, το λειτουργικό τμήμα, τότε η Επιτροπή μπορεί να αναθεωρήσει τη θέση της. Έχουμε ορισμένες ε, διαφάνειες. Έχετε ένα έγγραφο που σας ε, παραδώσαμε. Τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη περίοδο αναφόρας 2015-2019 έχουμε φτάσει σε ε, στόχους για την Ένωση ήδη το Μάρτιο του 2014 και τον Ιούλιο και το Μάρτιο του 2015 η Επιτροπή έλαβε απόφαση για τα σχέδια απόδοσης. Μερικά ε, συμμορφούνται προς τους στόχους, αλλά όμως ε, δεν συμμορφώνονται με τους στόχους και γι' αυτό αναθεωρούνται ορισμένα λειτουργικά τμήματα. Όλες αυτές τις πληροφορίες θα τις βρείτε στο έγγραφο που σας αποστήλαμε. Για αυτούς που δεν συμμορφώνονται θα πρέπει να αναθεωρήσουν το σχέδιο απόβασης και η Επιτροπή έλαβε μία απόφαση το Φεβρουάριο του 2016 ε, η απόφαση ήταν θετική για ορισμένα λειτουργικά τμήματα, για ορισμένα όμως ε, τμήματα η απόφαση είναι αρνητική σε σχέση με την ε, αποδοτικότητα του κόστους. Ε, σε σχέση με την Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα ως προς τις ικανότητες η απόφαση είναι αρνητική επί του παρόντος. Βρισκόμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη. Στην Επιτροπή ε, του Ενιαίου Ουρανού θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια τελική επίλυση του ζητήματος και με τα σώματα αναθεώρησης ε, δεδομένων, ιδιαίτερα για την Κύπρο και την Ελλάδα, όπου, υπάρχει διαρθρωτική, όπου υπάρχουν διαρθρωτικές ε, καθυστερήσεις και υπάρχουν προβλήματα και με τη Γαλλία σε σχέση με τα κέντρα ελέγχου εναέριας ε, κυκλοφορίας. και που δημιουργούν καθυστερήσεις. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα σε σχέση με την αποδοτικότητα της ΦΑΜΠΕ και αυτό οφείλεται σε πολύ ψηλό κόστος αναμονάδα στη Γερμανία. Και στη Γαλλία οι στόχοι απόδοσης ε, δεν ε, συμβαδίζουν με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Είχαμε και την υποστήριξη ενός σώματος ε, αποτίμησης αποδόσεων και προσπαθήσαμε να δούμε κατά πόσο υπάρχει πραγματική απόδοση και αποδοτικότητα ανάλογα με τα σχέδια αυτά και την εφαρμογή τους. Η δημιουργία ενός FAB έχει μείνει πίσω και γι' αυτό τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να μεταφέρουν αυτή την ενιολογική βάση στον, ε, την ε, νομοθεσία τους για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Φέτος είδαμε μετά το 2012 που ήταν ε, η ημερομηνία ορόσημο για την εφαρμογή των σχεδίων, είδαμε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος θεσμικά μέσα στα πλαίσια των ΦΑΜΠ αλλά ε, δυστυχώς δεν φτάσαμε σε αυτά ευεργετήματα σε σχέση με την χρήση του εναέριου χώρου και τελικά και για τους επιβάτες. Η Επιτροπή αποφάσισε ε, φέτος να ανοίξει μια διαδικασία ε, παραβάσεων ενώπιον του δικαστηρίου για να δούμε ποιο είναι το λειτουργικό ευεργέτημα που απορρέει από αυτές τις επιμέρους χρήσεις. Μετά το 2012 έτσι η Επιτροπή θα μπορέσει να κρίνει καλύτερα εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Εμείς θεωρούμε ότι δεν επαρκούν. Θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση και εάν η έννοια του ΦΑΜΠ ισχύει, μπορεί να ισχύει και για το μέλλον, τότε θα δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. για να υπάρχει μία σωστή διαχείριση του εναέριου χώρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βιμ Φαντεκάμπ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να ομολογήσω πως δεν είμαι ειδικό στο θέμα. Αυτό θα περιοριστώ σε δύο ερωτήματα. Αυτό το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ και μετά από αυτά τα οποία μας είπε η Κομισιόν είναι είμαστε ικανοποιημένοι ή όχι τώρα. Τε, τα έκαναν καλά τα κράτη-μέλη ή όχι. Γιατί δεν μπορώ εγώ να τα κρίνω αυτά τα πολιτικά. Τα... Δεν μπορώ να κρίνω, με πολιτικά το ζήτημα. Ή ε, καθυστερήσαμε όπως συνηθίζουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη ερώτηση. Τι θα συμβεί από εδώ και Έχουμε το 6 συν 2. Ε, ποια είναι λοιπόν τα επόμενα βήματα, πώς το βλέπει η Κομισιόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και εγώ. Ισμαήλ Ερτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Θεωρώ πως η ουσία είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φαντεκάμπ. Κοιτάξτε, δεν είναι δικιά μας ε, δικό μας το θέμα. Τα κράτη-μέλη εδώ πέρα δεν συμφωνούν και θα ήθελα να ακούσω τι άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι, τι σκοπεύει να κάνει για να κινητοποιηθούν. Γιατί αυτά τα οποία έχουν υποβληθεί Εντάξει, εμένα κάπως ε, με διευθύνουν, αλλά λένε πώς θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο για το πώς θα συνεισφέρουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κατάλαβα καλά, θα υπάρξει μια ε, αξιολόγηση των κρατών μελών για το εάν τηρούν τις προδιαγραφές ή όχι. Δεν ξέρω, είναι τόσο εύκολο να κρίνουμε την απόδοση των άλλων χωρίς προβλήματα. Και το δεύτερο μου ερώτημα. Μήπως υπάρχει κάποια καλύτερη λύση για να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να φτιάξουν επιτέλους αυτά τα μπλοκ αέριου χώρου. Ευχαριστώ, Τζάκι Πόστερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και οφείλω να πω πως εκπλήσωνα από αυτά τα οποία μας λέει η Κομισιόν. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν εδώ πέρα στην πρώτη μου εντολή όταν αρχίσαμε να μιλάμε για τον ενίο ευρωπαϊκό νερό. Πριν από 10 χρόνια, στην προηγούμενη μου θητεία, ήμουν εισηγήτρια για να ξεκινήσει η υπόθεση αυτή. Πριν αρχίσουμε να συζητάμε καν το ΣΕΖΑΡ, το 2 και όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να συνυπογράψουν τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Κοιτάξτε, δεν είμαστε αφελείς, ε, γνωρίζουμε πως υπάρχουν προκλήσεις και δυσκολίες ε, όταν έχουμε ένα τόσο δύσκολο θέμα. Αλλά όταν κοιτάμε τα θετικά και ανέφερε ήδη ο πρόεδρος ε, κάποια πράγματα, π.χ. απευθείας δρομολόγια Ε, λιγότερα καύσιμα. Και για όλα αυτά τα πράγματα ήταν σαφές πριν από 12 χρόνια γιατί ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και ακόμα και εγώ ως συντηρητικός ε, είχα αναγνωρίσει πως δεν ήταν θέμα κυριαρχίας. Ε, πάντα τα κράτη-μέλη θα ελέγχουν τον ένα χώρο τους. Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε ήταν να προχωρήσει αυτό το θέμα και είχαμε την πρόταση, την ε, συλλογική πρόταση να περάσουμε σε μια αναδιάρθρωση ονόματι FABS. Κάποια κρατημέλη έχουν ήδη συμμορφωθεί. Ηνωμένο Βασίλειο, Σκανδιναβία. Είμαστε το 2016, ήμουν στην Κύπρο. Ε, όταν η Κύπρος και η Ελλάδα συνυπέγραψαν για το δικό τους το FAB. Και αυτό ήταν πάρει στην προηγούμενη θητεία, 2013-2014. Και σήμερα έρχεστε ε, και μας λέτε, ε, όχι εσείς προσωπικά δηλαδή, με κομισιόν, μας λέτε για όλα αυτά τα σχέδια της ε, απόδοσης. Δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να προχωρήσουμε, να ασχοληθούμε με την ουσία αυτό το οποίο δεν κάνετε εσείς ως Κομισιόν είναι να πιέζετε τα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται και δεν δημιουργούν τα φαμπ τα οποία απαιτούνται για να έχουμε μετά μια πραγματικά κοινή διαδικασία για να ξεκινήσει το ΣΕΖΑΡ. Δεν είναι λοιπόν έκθεση αυτό το οποίο μας κάνετε. Τι είναι άλλες ε, εφαρμοστικές πράξεις, ε, κάποια εφαρμοστικά μέτρα. Να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση και αυτό αντιμετωπίζεται γιατί δεν βοηθάν τα κράτη-μέλη, αν δείτε τους παρόχους και τις ε, κυβερνήσεις που δεν κάνουν τίποτα για να το προωθήσουν το θέμα. Αλλά αυτό είναι αδιάφορο. Αδιάφορο. Δεν μπορεί να έχουμε μια κατάσταση αμοιβαία υποφελή εάν δεν συμμορφωνται καποια κάποια κράτη-μέλη. Η δικιά σας η δουλειά λοιπόν ως Κομισιόν η αστυνομία αν θέλετε εδώ πέρα να ε, προχωρήσετε το θέμα και ειλικρινά δεν ε, κάνετε εδώ πέρα την δουλειά σας επαρκώς τουλάχιστον για τη δική μου την ε, ομάδα και την Επιτροπή νομίζω. Λοιπόν, προτείνω. Φύγετε από εδώ σήμερα και όταν ξανάρθετε δώστε μας μια σωστή ενημέρωση για το που βρίσκονται τα FAB. Τώρα αυτά εδώ πέρα που μας λέτε πόσα ευρώ κοστίζει και τα λοιπά τα ξέρουμε. Γι' αυτό είμαι σε αυτή την Επιτροπή. Και το καταλαβαίνουν και τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Απαντήσεις δεν έχουμε. Προχωράμε καθόλου. Από ό,τι βλέπω, όχι. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να έρθει το συντομότερο δυνατόν και να μας δώσει μια σωστή ενημέρωση. Πού είναι οι καθυστερήσεις, πού είναι η στενοποίοι, γιατί θέλω να ξέρω ποια κράτη-μέλη μπλοκάρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Γκεζίνε Να συμφωνήσω. Ε, ε χρόνια το συζητούμε αυτόν τον ενιαίο ουρανό. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να ασχοληθούμε με την ουσία επιτέλους. Μας απασχολεί όλου. Πολλέ φορές έχω πει ότι αν ήξεραν όλοι οι ε, πολίτες ε, πόσο, με πόσο μη βιώσιμο τρόπο διαχειριζόμαστε τον ενιαίο ουρανό μας, Πραγματικά θα... Δεν ξέρω τι θα έλεγαν. Είναι τεράστια τα κόστη που υπάρχουν, οι καθυστερήσει, ε, οι... χάνουν και οι πολίτε, χάνουν και οι αεροπορικέ εταιρείε. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε μια λύση. Τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι έτοιμα να κάνουν πραγματικά αυτό που έχουν υπογράψει ότι θα κάνουν. Γιατί όλοι λέμε ότι το χρειαζόμαστε. Όλοι συμφωνούμε. Και τελικά αρνούνται τα κράτη-μέλη να το εφαρμόσουν. Και βεβαίω ουσιαστικά η Κομισιόν πρέπει να δει τι θα κάνει. Η Κομισιόν ουσιαστικά είναι η, ε, η υπεύθυνη για να διαφυλάξει τις, ε, τις συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να ε, ασχοληθεί και να φέρει τα κράτη-μέλη στο σωστό δρόμο. Έχουμε και το θέμα του Γιβραλτάρ. Μιλάμε για την κινητικότητα εντός της Ευρώπης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε να την εξασφαλίσουμε και για, τον, για τις ενέργειες της Θέλουμε να λύσουμε και τα θέματα μεταφορών, κινητικότητα. Η Κομισιόν λοιπόν πρέπει να έχει μια παρόμοια προσέγγιση. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσουμε, αλλά Αναρωτιόμαι, υπάρχει κάποια δυνατότητα η Κομισιόν να έχει πιο σκληρή στάση. Και τώρα έχω ένα ερώτημα για αυτό που είπατε συγκεκριμένα. Είπατε στην αρχή ότι η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν προβλήματα δυνατοτήτων υποδομών. Το έχω ακούσει και εγώ, ότι είναι δύσκολο στην Ελλάδα, ας πούμε, να προσγειωθεί κανείς ή ότι ε, θα μπορούσε ίσως να υπάρχουν περισσότερες πτήσει προς την Ελλάδα ή προς την Κύπρο, ότι υπάρχουν προβλήματα υποδομών. Θα ήθελα από εσά να μου πείτε ποια είναι τα προβλήματα αυτά υποδομών. Δεν υπάρχουν ε, καταρτισμένο προσωπικό, τι λείπει και τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να το αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι σημαντικό για τις χώρες να ε, αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Είναι ε, ελκυστικοί προορισμοί για διακοπές, πάνε πολύ Οπότε καλό θα ήταν να λυθούν τα προβλήματα αυτά γιατί η κατάσταση προφανώ δεν θα είναι πολύ καλή. Επίση, για αυτό τον πίνακα που κάνατε, αναρωτιέμαι. Όταν ε, όταν ξεκίνησαν να εφαρμόζονται αυτά τα FABs για μικρές χώρες όπως η Ελβετία ή το Λουξεμβούργο ήταν έτοιμα να παρέμβουν, να δράσουν ίσως περισσότερο από μεγαλύτερες χώρες και τώρα βλέπουμε αυτό το, το, πίνακα για την αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τη, το κόστος. Η Γερμανία πάει καλά από ό,τι βλέπω και πραγματικά με εκπλήσει αυτό γιατί Νόμιζα ότι είχε μείνει λίγο πίσω η Γερμανία ως προς αυτό. Οι κάτω χώρες, Βέλγιο και Λουξεμβούργο ε, δεν πάνε τόσο καλά, οπότε δεν καταλαβαίνω ακριβώς πώς το αξιολογήσατε αυτό. Και η Γαλλία εξίσου άσχημα. Μείον 4,1, μείον 4,5 είναι, όπως οι χώρες Μπενελούξ. Ε, για τη Γαλλία, με τι σχετίζεται αυτό, ότι είχαν πολλές απεργίες, ας πούμε, ότι δεν ε, πραγματοποιήθηκαν κάποιες πτήσεις όπως είχαν προγραμματιστεί. Για ποιο λόγο έχετε καταλήξει αυτή την αξιολόγηση του τον πίνακα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλοι συμφωνούμε και λέμε το εξής. Πώς ο κανονισμός του ενιαίου ουρανού είναι πολύ καλή πρωτοβουλία του 2004, μετά αναθεωρήθηκε το 9 και μετά ε, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2012. Αυτό αναφέρεται. Σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Είπατε ότι ναι, υπάρχει ευθύνη των κρατών, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ ο Ευρωπαϊκός Ενιαίος ε, Ουρανός. Γιατί μπορούμε να συνεργαστούμε για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα θα πρέπει εντάχει να βρούμε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να κινηθούν κάπως. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε, έχετε αποτελέσματα από πλευράς περιβάλλοντος για τα δύο λειτουργικά τμήματα που είναι πιο προχωρημένα, ε, Μπενελούξ, ε, Γαλλία, ε, Γερμανία και το δεύτερο μπλοκ που αφορά τις ανατολικές χώρες. Έχετε δει επίσης ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω και εγώ. Κοιτάξτε, ε, γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται με τους εθνικούς εγωισμούς, αλλά εδώ πέρα βλάπτει και τα εθνικά συμφέροντα. Γιατί, πρώτα απ' όλα, ε, υπάρχει περισσότερη ασφάλεια. Ε, αυτό θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει όλους. Να είναι ως δυνατόν μεγαλύτερη ασφαλεία. Δεν συμβαίνει. Δεύτερον, εξοικονομούμε χρήματα. Αν έχουμε παντού αυτά τα θεσμικά όργανα. Κοστίζει αυτό. Προφανώς τα κάτι μέλη είναι τόσο πλούσια που αδιαφορούν. Δηλαδή μπορούν να εξοικονομήσουν λεφτά και εκπομπέ, αλλα αλλά κάποια κράτη-μέλη δίνουν δισεκατομμύρια για να περιορίσουν τις εκπομπές κατά 1-2%. Και εδώ πέρα μπορούν να εξοικονομήσουν λεφτά και δεν κάνουν τίποτα. Ε, δεν είναι δυνατόν αλλά η Τζάκι Φώστερ είπε ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης. Μα αυτό υπάρχει και στην Κομισιόν. Και εγώ παρακολουθώ την υπόθεση αυτή 12 χρόνια. Και επί Γιαρζεμπόσκη, επί έκθεση Γιαρζεμπόφσκι το έχουν πει. Γιατί δεν συμβαίνει τίποτα. Έχουν υπογράψει τι συνθήκες, υποτίθεται ότι είμαστε ένα σύστημα δικαίου. Υπάρχει αν αρνούνται τα κράτη-μέλη να το κάνουν ο θεματοφύλακας των συνθήκων, δηλαδή η Κομισιόν. Γιατί δεν λέτε ε, ότι πρέπει να ξεκινήσει ή έχουμε ξεκινήσει διαδικασία παραβάση κατά των χ ωμέγα χωρών. Γιατί και με την ε, παραβίαση αυτή ε, μειώνεται η ασφάλεια, αυξάνονται οι εκπομπές και εξοδεύουμε και χρήματα στην Ευρώπη. Θέμε να ξέρουμε, καλά δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ, αλλά θέμε να ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης δεν υπάρχει μόνο στα κράτη-μέλη, αλλά από ό,τι φαίνεται και στην Κομισιόν. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα, τι θα κάνει η Επίτροπος. Ξέρω πως στην ιεραρχία, οι Επίτροποι, ε, εντάξει, ίσως να μπορούν να κάνουν και πολλά. Ο κύριος Τίμερμανς λοιπόν μας λέει συνεχώς better regulation. Ορίστε, εδώ πέρα λοιπόν τι έχουμε. Κακή ρύθμιση. Τι συμβαίνει. Θέλω κάποια απάντηση. Τα ξέρουμε τα προβλήματα, τα έχουμε ακούσει 100 φορές. Ή πείτε μας τουλάχιστον τι κάνατε εσείς αφού δεν γίνεται τίποτα. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Λοιπόν, έχετε το λόγο και περιμένω να ακούσω τι θα μας πείτε. Okay. Thank you. Thank you, Uh, so... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ξεκινώντας από τον κύριο Κάμπ, μας ρώτησε κατά πόσο είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχει πρόβλημα με το μικρόφωνο. Direct in, then it is louder. If you make it so, it is not so loud. Yeah, sorry. Sorry, I start again. Θα ξαναρχίσω. Ε, θα ε, αρχίσω από την ερώτηση του κυρίου Βάντερ Κάμπ. Κατά πόσο είμαστε ικανοποιημένοι, ρώτησε, με την εφαρμογή των ΦΑΜΠ». Όχι, φυσικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί αρχικά αυτά που προβλέπονταν από την ομοθεσία δεν τηρήθηκαν. Πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία και φυσικά τα κράτη-μέλη λένε ότι σε αυτό το τομέα δεν μπορούμε ε, να έχουμε γρήγορες αλλαγές. Όλα θα πρέπει να γίνουν βαθμιαία. Και μιλήσατε για το τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα αντιδράσουμε, ποια θα είναι τα μελλοντικά βήματα. Ως προς τα FAB δυστυχώς ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία στον ε, ε, ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Προσπαθούμε να προωθήσουμε το ΣΕΖΑΡ καταρχήν που είναι ο τεχνολογικός ε, πυλώνας στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο για να προβούμε στη συνέχεια και στις τεχνικές αλλαγές, ε, δηλαδή την, ε, ε, στο θέμα της πλοήγησης και ούτω καθεξής, δηλαδή θέματα στα οποία μπορεί να μας βοηθήσει το ΣΕΖΑΡ. Αλλά όχι τα ίδια τα ΦΑΜ, δεν μας ικανοποιούν. Επίσης, έγινε λόγος για το σχέδιο απόδοσης για τους στόχους. Το σχέδιο απόδοσης εισήχθη για να γίνουν αλλαγές, έτσι δηλαδή ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών ε, πλοήγησης να μας δώσουν νέα στοιχεία πιο αποδοτικά. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμα τα κράτη-μέλη αντιστέκονται. Όχι όλα, αλλά πολλά από αυτά. Και τα κράτη-μέλη είναι αλληλέγγυα μεταξύ τους, δεν θέλουν να στραφούν το ένα κατά του άλλου και ε, γι' αυτό αυτή η αρχή της αλληλεγγύης μας αποτρέπει από το να φτάσουμε σε αποτελέσματα. Ε, κύριε Φώστερ, κατανοώ την αντίδρασή σας, αλλά το θέμα ε, της ημερήσιας διάταξης αφορούσε τα σχέδια απόδοσης. Υπάρχουν μερικά FAB που έχουν ε, προχωρήσει αρκετά όπως το δανέζικο και το σουηδικό. Ίσως υπάρχει έλλειψη πολιτικής θέλησης. Δεν είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, αλλά εθνικού συμφέροντος και υπάρχουν και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Μετά το καλοκαίρι θα σας δώσουμε μία πλήρη επισκόπηση για το που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτά τα λειτουργικά τμήματα του Ευρωπαϊκού Εναερίου Χώρου. Η κυρία Μάισνερ είπε ότι εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες των ε, συνθήκων. Έχουμε ξεκινήσει ε, τις ε, προσφυγές κατά των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τα FAB. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση επιστολών όχλησης και στη Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία και Μπενελούξ ε, έχουμε ζητήσει αιτιολογημένες επεξηγήσεις σε σχέση με την εφαρμογή των FAB. Έχουμε ξεκινήσει τις ε, διαδικασίες προσφυγών. Αναφερθήκατε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ναι, το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη ελέγχου. Μάλλον η έλλειψη προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Σε ορισμένα κράτη-μέλη ισχύει αυτό, ιδιαίτερα σε ώρες εχμής. Δηλαδή, πολλές, ε, ε πολλοί ελεγκτές στη Γαλλία ε, δεν επιθυμούν να προσέλθουν στην εργασία τόσο νωρίς το πρωί. Υπάρχουν δηλαδή και θέματα ε, κοινωνικών διεκδικήσεων και αναταραχών και γι' αυτό έχει σημασία και το ωράριο εργασίας των ε, ελεγκτών ενέργειας ε, κυκλοφορίας, δηλαδή η διαθεσιμότητα της ώρες εχμής το καλοκαίρι και της περιόδους εχμής. Ο κύριος Ντέλη Ε, μίλησε για νέα μέτρα, σας είπα ότι το ΣΕΖΑΡ είναι η καλύτερη λύση για τον εξυγχρονισμό του, των συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας σε σχέση με τα αποτελέσματα ε, και τις επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος με το ΣΕΖΑΡ τώρα υπάρχει ε, αποδότη, υπάρχει απόδοση κατά την πτήση, ενεργειακή απόδοση και με αυτά τα μπλοκ ελέγχουμε και τις επιπτώσεις ε, επί του περιβάλλοντος. Και γίνονται πολλές εξοικονομήσεις ως προς τα καύσιμα και οι επιπτώσεις ε, των πτήσεων κατά του περιβάλλοντος περιορίζονται. Άρα επιτελείται πραγματικά πρόοδος. Τέλος, σε σχέση με τα σχόλια του Προέδρου ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής θέλησης στα κράτη-μέλη και κατά πόσο η Επίτροπη μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, βεβαίως και μπορούμε, Γι' αυτό αρχίσαμε και με τις προσφυγές κατά των κρατών μελών. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και να επιμείνουμε. Αυτό το συζητάμε ήδη. Βεβαίως κατά την ε, ψηφοφορία έχουμε ε, την αντίσταση των κρατών μελών αλλά αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2000, έγινε πραγματικότητα το 2004 ε, επί, της, ε, επί της Επιτροπής Λογιόλαντε Παλάσιο. Έκτοτε όμως άλλαξε η κατάσταση γιατί επήλθε η μεγάλη οικονομική κρίση το 2007 2008 και μιλάμε όχι τόσο για ικανότητα, αλλά για αποδο... οικονομική απόδοση γιατί υπήρξαν μεγάλες αλλαγές και μειώσεις πτήσεων. Το σύστημα είναι κατακαιρματισμένο ακόμα, μην το ξεχνάτε. και αν αντιμετωπίσουμε άλλη μία κρίση, το σύστημα δεν θα είναι πια ε, βιώσιμο. Υπάρχουν ανάμεικτα αποτελέσματα ως προς την τεχνολογική πρόοδο, ε, την εφαρμόζουμε, αλλά από θεσμικής και οργανωτικής πλευράς για την ε, συγχώνευση κέντρων εναέριας κυκλοφορίας. Δυστυχώς ε, έχουμε μείνει πίσω γιατί υπάρχει θέμα εθνική, εθνικού συμφέροντος. Κάθε κράτος θέλει για λόγους γοήτρου, ε, κυριαρχίας να κρατήσει το δικό του κέντρο εναέριας κυκλοφορίας. Δηλαδή, ε, στα λόγια λένε ναι, αλλά έμπρακτα δεν ακολουθούν. Άρα δεν είναι καθόλου εύκολο για μας. Ευχαριστώ. Κανένας όμως δεν είναι ευχαριστημένος, θα το καταλάβατε φαντάζομαι. Δώδεκα χρόνια την ε, παλεύουμε αυτή την νομοθεσία και έχουμε και τα τελευταία χρόνια για την, της οικονομικής ε, κρίσης, γιατί όλα τα παράπονα ενισχύθηκαν, χάνουμε λεφτά. Ε, Όλοι τα ξέρουμε τα επιχειρήματα των κρατών μελών, αλλά εσείς γιατί δεν μπορείτε να, να ξεκινήσετε μια νομική δράση, κάτι. Ε, χρόνια το ζητάμε, γιατί δεν γίνεται τελικά. Ποιος είναι αυτός ο λόγος που η Κομισιόν σε αυτό το σημείο δεν δρά ως θεματοφύλακα των συνθήκων και να πει πρέπει να το κάνετε. Το έχετε υπογράψει, πρέπει να τηρήσετε την υπογραφή σας. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει από την προς. Ξέρω ότι εσείς ε, μας ε, ενημερώνετε για το τι γίνεται και ξέρετε την κατάσταση, αλλά καλό θα ήταν ίσως να μας κάνετε τη χάρη να πάτε και λίγο πιο ψηλά στην ιεραρχία και με κάποιο τρόπο να προχωρήσει το πράγμα, γιατί όπως καταλάβατε από όλους μας δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Να γνωρίζουμε ότι είσαστε σε δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού ελεγκτών. Το να κάθεστε και να λέτε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν προβλήματα. Ε, μιλάμε για περιόδους εχμής. Ο οποιοδήποτε ελεγκτής ή πιλότος ότι όταν δέχονται ένα συμβόλαιο είναι μία εργασία 24 ώρες 7 ημέρες της εβδομάδας. Άρα τη στιγμή που οι πολιτικοί δεν μπορούν να δεχτούν αυτές τις προκλήσεις, μα αυτό δεν αρκεί. Ο πρόεδρος ήταν σαφής. Γιατί δεν προωθείτε μια διαδικασία επί παραβάση άμεσα. Δηλαδή, αν δείτε τη Γαλλία, την Ισπανία, πρόκειται για κομβικά σημεία και το ξέρετε. Εσείς δεν προχωράτε Υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, αλλά μη μας λέτε τώρα ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, γιατί αλλού λειτουργεί πολύ καλά το σύστημα. Εμείς μιλάμε και με το Συμβούλιο δεν είναι απάντηση το να μας λέτε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, γιατί δεν είναι αυτή η αιτία του κακού. Ευχαριστούμε. Αν θέλετε να ξαναπάρετε το λόγο, Κομισιόν, ευχαριστώ. Ναι, σύντομα. Για, το, ε, για την έλλειψη ελεγκτών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα στην Ελλάδα σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των ελεγκτών. Πρέπει να ανοίξουν λοιπόν νέοι τομεί. Ε, και έγινε μια προσφορά από την Ιταλία να σταλεί μια ομάδα ελεγκτών, 20 νομίζω, στην Ελλάδα, και αυτή η, αυτή η πρόταση απερίφθη. Γιατί, γιατί οι ελεγκτέ πρέπει να είναι Έλληνε, να μιλάνε ελληνικά. Καταλαβαίνετε. Μπορεί να μην υπάρχει έλλειψη αν δείτε συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ελεγκτέ, αλλά αν δείτε σε τοπικό επίπεδο, σε κρατικό, υπάρχει έλλειψη. Υπάρχουν χώρε που έχουν πολλού ελεγκτέ, όπω η Γερμανία α πούμε, έχουν ε, πλεόνασμα ελεγκτών. Αλλά το να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι ελεγκτέ σε άλλε χώρε είναι αδύνατο σχεδόν. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ. Ωραία. Οπότε. Κανένα δεν είναι ευχαριστημένο, το διαπιστώνουμε όλοι, αλλά όλοι τουλάχιστον είμαστε αισιόδοξοι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το υγρό ποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση αερίου. Ε, Κλάουντια Μοντέιρο είναι η συγγήτρια. Έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι αυτή η γνωμοδότηση εντάσσεται στο θέμα της ενεργειακής και βιώσιμης ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποθήκευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο λοιπόν το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά ε, καύσιμα και το οποίο έχει θετικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δηλαδή ε, δεν ε, έχει τόσο υψηλές εκπομπές και δεν πλήττει το περιβάλλον. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο εγγυάται την ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση με τη γνωμοδότηση αυτή άκουσα διάφορες οργανώσεις, επιχειρήσεις του τομέα που μας είπαν πώς έχει κατάσταση ως προς το υγροποιημένο αέριο στα κράτη-μέλη. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στις ε, θαλάσσιες μεταφορές έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος των εκπομπών και θα χρησιμοποιείται από όλα τα πλοία τα οποία ελιμενίζονται σε ευρωπαϊκούς λιμένες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ο νομοθέτης θα πρέπει να ορίσει ορισμένες προτεραιότητες. Θα πρέπει στα κοινοτικά λιμάνια να ορίσουμε τις ε, ασφαλείς συνθήκες χρήσης και μεταφοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μπορείτε να, μπορεί να χρησιμοποιείτε και στις ε, δημόσιες μεταφορές και για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Βεβαίως πάντα υπάρχουν κίνδυνοι τους οποίους θα πρέπει να αποτιμήσουμε και να αντισταθμίσουμε. Να μην υπάρχει διαρροή μεθανίου πρωτίστως και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα τεχνολογικά μέσα εχμής για να ανταποκριθούμε. Μέσα τα οποία είναι ε, διαθέσιμα για να μην έχουμε συγκεκριμένες αρνητικές απόρριες. Θα ήθελα να αναφερθώ και στο θέμα των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών. Η οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα ε, μιλά για ένα πλαίσιο εφαρμογής μέχρι τον Νοέμβριο του 2017. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα μικρά λιμάνια και εσωτερικά λιμάνια προμήθειας ε, υγρού φυσικού αερίου. Τώρα, η αγορά αφορά και τα δίκτυα διανομής. Δεν έχουμε τερματικούς σταθμούς παντού δεν είναι ίση η κατανομή τους και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή, αυτό τον κατακαιρματισμό. Όλα τα λιμάνια θα πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτή τη δραστηριότητα μέσω ΣΕΦ. συνδέοντας την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να προσδώσουμε μεγάλη ε, σημασία στα απομακρυσμένα λιμάνια όταν μιλάμε για εγκατάσταση τερματικών σταθμών και δίκτυα παροχής. Ένα άλλο θέμα αφορά τις επενδύσεις. Η Επιτροπή μας μίλησε για τις δικές εναλλακτικές ε, λύσεις σε σχέση με την αποθήκευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Υπάρχει ένας ενδυνάμει αγωγός στη Μαδέρα, καθώς και λιμάνια δορυφόρη. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη η κατασκευή τερματικών σταθμών. Υπάρχουν όμως δυνατότητες και ευκαιρίες, τις οποίες δεν πρέπει να χάσουμε. Ελπίζουμε η στρατηγική αυτή να μην, να μην δημιουργήσει περισσότερα, ε, περισσότερες, ε, ε, περισσότερους ενεργειακούς θύλακες από αυτούς που χρειάζονται. Η Ευρώπη διαθέτει υψηλό αριθμό τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Δεν είναι θέμα του παρόντος. Έχουμε 1.500 φορτηγά που κινούνται και με υγροποιημένο και έχουμε ένα υψηλό αριθμό πλοίων παγκοσμίω που κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θα πρέπει να έχουμε με ένα ευρύ φάσμα ε, χρήσης αυτού του, αυτής της μορφής του αερίου υπάρχουν και περιορισμοί. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να επεκταθώ περισσότερο. Είμαι στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε για οποιασδήποτε τροπολογίες. Να το δούμε μαζί με τους σκιώδεις για να φτάσουμε σε ένα συνενετικό και σαφές έγγραφο το οποίο να μην προβαίνει σε αποκλισμούς, αλλά να επιτρέπει την ευρύτερη χρήση του υγροποιημένου ε, φυσικού αερίου για ένα τομέα που είναι τόσο σημαντικό για εμάς, το τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ, Τερέζα Γκρίφιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κύριε εισηγήτρια, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για το πρώτο αυτό θετικό σχέδιο και το πώς δουλέψατε. Υποστηρίζω πάρα πολλές πτυχές και θετικές και αναφορές σε ΑΠΕ και εναλλακτικά καύσιμα για το LNG στις μεταφορές πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό καύσιμο, ειδικά όταν αντικαθιστά πιο ρηπογόνα συμβατικά καύσιμα και δεν υποκαθιστά απε, ειδικά στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών όμως πρέπει τα κράτη-μέλη ενώ αναπτύσσουν ε, την υποδομή τους, να αξιολογήσουν σωστά την ζήτηση του φυσικού αερίου για να μην έχουμε κάποια κάποιες υποδομές αποκλεισμένες. Επίσης, οι νέες αυτές οι υποδομές δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουν την αποκλειστική υιοθέτηση μιας τεχνολογίας, ειδικά ορυκτών καυσίμων. Πρέπει να προωθήσουμε την χρήση υφιστάμενων τέρμιναλ μαζί με την ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς αερίου με διασυνδέσεις. Και τέλος και πιο σημαντικό, πρέπει να διασφαλίσουμε πως ε, οι στόχοι ΑΠΕ και αποτελεσματική χρήση ενέργεια θα πηγαίνουν χέρι-χέρι με την χρήση και ανάπτυξη φυσικού αερίου. Δεν μπορεί το υγροποιημένο φυσικό αέριο να υπονομεύσει την ανάγκη να απομακρυνθούμε από τον άνθρακα ούτε να αποτελέσει την πίσω πόρτα του σχιστολιθικού αερίου. Πρόκειται λοιπόν για μια μείωση απλά η οποία από μόνη της δεν είναι βιώσιμη. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε βιώσιμη την χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου και να τηρηθεί η πολιτική των ΑΠΕ. Και αναμένουμε και τη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ρόμπερτ Τσίλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Τόμας Παραγκαχ είναι σκιοδησηγητής, θα μεταφέρω τα λόγια του. Θεωρούμε πως ε, η στρατηγική αυτή είναι σημαντικό κομμάτι ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Σημειώνουμε πως ε, τα τέρμιναλ αποτελούν σημαντικό κομμάτι της επαναεριοποίησης, όμως χρησιμοποιούνται μόνο κατά 20%. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια υποδομή διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Επίσης, καλοδεχούμενη ιδέα Αύξηση ε, των περιφερειακών συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσει σε καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αναγνωρίζουμε πως ο κανονισμός των Ευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας ε, μας δίνει το κατάλληλο πλαίσιο για να στηρίξουμε τις υποδομές του αερίου και βεβαίως τα τέρμιναλ μετάδοσης ε, και αποθήκευσης. Το ECR επίσης θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και να έχουν όλα τα κράτη-μέλη πρόσβαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτή είναι η άποψή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γιώζο Ράντος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Άλντε να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Μοντέιρο Ντεαγιάρ για την στρατηγική στήριξη του υγροποιημένου φυσικού αερίου το οποίο θα υποκαταστήσει πιο ρηπογόνα καύσιμα. Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα που θεωρώ πως πρέπει να υποθούν. Πρώτα απ' όλα στη γενική έκθεση νομίζω πως είναι σημαντικό να τονίσουμε την ε, έγκριση έργων κοινού ενδιαφέροντος γιατί βεβαίως αυτό έχει μεγάλη σημασία για να ωφεληθούν όλα τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, αυτό σχετίζεται με την γνωμοδότησή μας. Νομίζω στην γνωμοδότηση της Επιτροπής μας μιλάμε για την κατασκευή των σημείων LNG ειδικά στα λιμάνια εκείνα τα οποία δεν είναι στο δίκτυο πυρήνα των διευρωπαϊκών δικτύων ε, μεταφορών. Αυτό νομίζω αφορά ιδιαίτερως την Επιτροπή μας. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μαρία Κίλεν. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω ε, την συγγετρία γιατί ήταν ε, πολύ καλή η έκθεσή της βασίζεται σε εμπειρογνωμοσύνη, είναι ισόρροπη. Θα υποβάλουμε κάποιες προτάσεις βεβαίως εμείς ε, για κάποιες τροπολογίες. Ε, για, το, την περίοδο μετά το ε, LNG. Αν έχω καταλάβει καλά, το Κοινοβούλιο έχει μια κοινή ενιαία άποψη για την σημασία του LNG ως α, καύσιμο για μια μεταβατική περίοδο, αλλά για μετά από αυτό πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ενεργειακή διαθεσιμότητα και ε, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη και την παραγωγή ε, LBG και τήρηση των ε, προϋποθέσεων που υπάρχουν για την διανομή. Νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στην έκθεση. Επίσης, σε σχέση με αυτό, είναι απαραίτητο να δώσουμε προσοχή στα κίνητρα προς τους ε, operators ε, υγροποιημένου αερίου. Και επίσης ε, πρέπει να δούμε τον εξοχρονισμό των σαφών, βεβαίως και την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και θέλω έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια γιατί έκανε μια πολύ καλή αρχή. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανεί, ότι το LNG έχει καλύτερη απόδοση ό,τι αφορά το άζωτο και το θείο και τις εκπομπές οξυδίων αζώτου και θείου. αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ευαγγελική η προσέγγιση στην έκθεση, στην στήριξη που δίνει στο LNG. Και θα ήθελα εδώ να είμαστε λίγο προσεκτικοί γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες ε, ε, συνέπειες ε, αθέλητες για τις συστάσεις ας πούμε φορολόγησης για το ντίζελ έναντι του πετρελαίου γιατί ήταν πιο αποτελεσματικό ό,τι αφορά τον άνθρακα. Δεν είχαμε φανταστεί ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα μόλυνσης του αέρα, ούτε όταν υιοθετήσαμε την πρόταση για τα βιοκαύσιμα είχαμε σκεφτεί ότι μπορεί να έχουν ε, επιπτώσεις στην ε, διαφοροποίηση της ε, χρήσης της γης από την παραγωγή τροφίμων στην χρήση τους μόνο για ως βοσκοτόπια. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να το δούμε υπό το ίδιο φως. Μιλούμε για ένα ορυκτό καύσιμο. Μπορεί να είναι μεταβατικό καύσιμο λοιπόν. Και εγώ θα ήθελα ως τμήμα αυτής της, αυτού του επένου του LNG, να δούμε και έναν ισολογισμό ας πούμε για το LNG σε σχέση με την απόδοσή του και το περιβάλλον και να το συγκρίνουμε με τον αντίστοιχο ισολογισμό που θα έχουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να δούμε ότι μιλάμε για μια τεράστια διαδικασία προσαρμογής των υποδομών για την προμήθεια του όγκου του LNG που αναφέρεται στην έκθεση. Και επίσης πρέπει να έχουμε να, έναν δείκτη για, τις, ε, για, τον, για το διοξείδιο του άφρικα. Στην έκθεση μιλάμε πολύ για το ότι το LNG μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ε, εκπομπών του, ε, του θερμοκηπίου, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι δυνητικό που μπορεί να είναι όντως πολύ σημαντικό γιατί μιλούμε για 86 φορές περισσότερο ε, το δυναμικό υπερθέρμανση του πλανήτη του διοξιδίου του άνθρακα και έχοντας υπόψη ότι οι ε, η μελλοντική ε, τροφοδοσία του LNG θα έρθει από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ. με αποτέλεσμα, που θα είναι αποτέλεσμα fracking, μιλούμε για νέους κινδύνους που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε μια πραγματική ισορροπία εδώ και να έχουμε και αυτόν, αυτήν ακριβώς την, αυτόν το συγκριτικό πίνακα πριν πέσουμε με τα μούτρα σε αυτό που θα μπορούσε ίσως να είναι το τρίτο μεγαλύτερο ενεργειακό λάθος. Ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much, um, Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, κυρία Μοντέιρο, κυρία Συγήτρια, αγαπητά μέλη, συμφωνούμε ότι ότι το αέριο είναι ένα μεταβατικό καύσιμο προς μία οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα σε σχέση με άλλα ορικά καύσιμα εμείς συμβαδίζουμε με τις στρατηγικές 2030 και 2050 για το κλίμα και την ενέργεια, αλλά υπάρχουν προκλήσεις για να αποφύγουμε τις διαρροές, όπως υπογράμμισαν τα μέλη. Αυτό μπορεί να επιληθεί με διεθνή διάλογο για να υπάρχει καλή ρύθμιση όσον αφορά την παραγωγή αερίου και η χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών. Οι διαρροές μπορούν να συμβούν ε, παντού, αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να αποφευχθεί αν δράσουμε σωστά. Σε σχέση με τη στρατηγική για το υγροποιημένο, θα πρέπει να κλείσουμε τα κενά έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε ε, ένα πλαίσιο το οποίο στη συνέχεια θα ε, εγκαταλείψουμε. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει πλέον κατακαιρματισμό στην εσωτερική αγορά, όλοι να έχουν πρόσβαση στο LNG και ε, περιοχές που δεν συνδέονται με το δίκτυο φυσικού αερίου που δεν θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο και υπάρχει μεγάλο δυναμικό για τα νησιά του Ατλαντικού ή της Μεσογείου που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Επίσης υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τις μεταφορές, για τις θαλάσσιες ε, μεταφορές και θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στους κυρίους Τρίκας και Σμιτ Πάουερ που θα μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Thank you very much, Mr. Moser. Thank you very much. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μοντέιρο Ντε Γκιγιάρ και όλα τα μέλη που εκφράστηκαν για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το φυσικό ε, αέριο θέλει να αντικαταστήσει τα βαρέα ε, πετρέλαια που χρησιμοποιούνται και το ντίζελ. Ο στόχος μας είναι η μείωση της χρήσης του άνθρακα. Και εδώ το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το βιομεθάνιο ή συνθετικό φυσικό αέριο, κάτι το οποίο θα συνεισφέρει στη μείωση χρήσης άνθρακα. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να τονίσω το παράδειγμα της Σουηδίας, όπου το 70% του βιομεθανίου χρησιμοποιείται ε, στη, για τις θαλάσσιες ε, μεταφορές. Ξέρουμε ότι θέλουμε να μειώσουμε τις ε, επιβαρύνουσες εκπομπές και το φυσικό αέριο είναι πολύ σημαντικό. Ήδη 20.000 ε, πόλεις χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο στα λεωφορεία. Προσπαθούμε να ελέγξουμε και τις εκπομπές ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά έχει γίνει μεγάλη πρόοδος από τους θερματικούς σταθμούς μέχρι την, τον τελικό χρήστη. Και βλέπουμε ότι ορισμένες αυτοκίνητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν νέα προαπαιτούμενα όπως η Volvo και ως προς το βιομεθάνιο θα πρέπει να ε, πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές πριν μπει στην αγορά. Ως προς την, τις υποδομές ξέρετε ότι το ε, εναλλακτικό, τα εναλλακτικά ε, μέσα επιβάλλουν στα κράτη-μέλη μέχρι τον Νοέμβριο φέτος να υποβάλουν τα σχέδιά τους δηλαδή πληροφορίες για, το, για τις ελάχιστες υποδομές, ε, για τα σημεία ανεφοδιασμού, ε, για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, τον, τους διάβλους, τους διαδρόμους TEN-T. Ποια θα είναι τα σημεία ανεφοδιασμού στις πόλεις και στα λιμάνια. Και αυτό δυνάμει του διαδρόμου τεντή. Επίσης, η Επιτροπή ε, υποστηρίζει τα κράτη-μέλη για επιπρόσθετες υποδομές μέσω του CEF, του Connecting Facility και η τελευταία δημοπράτηση έγινε το Φεβρουάριο και θέλουμε να έχουμε μία ελάχιστη υποδομή για να μπορέσουμε να έχουμε οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Ευχαριστώ. Προθεσμία για τις ε, τροπολογίες 21 ε, Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Κλείνουμε λοιπόν την ε, πρωινή μας συνεδρίαση και πάμε στους εισηγητές για τους, για τις τριμερείς, για τους τριμερείς διαλόγους η οποία όμως θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, οπότε όσοι δεν μπορούν να παραμείνουν, παρακαλώ να αποχωρήσουν από την αίθουσα.